Καλώς welcome. Um, uh, στη συνεδρίαση της Επιτροπής ε, ΕΚΟΝ. Νομίζω ότι έχουμε δύο πολύ ε, ενδιαφέροντα θέματα να συζητήσουμε. Θα εκμεταλλευτώ όλο το χρόνο του Προέδρου για να πω τα διάφορα συνηθισμένα και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι θα πρέπει να περάσουμε στα βασικά μας θέματα γιατί έχουμε και ομιλητές. Όπως γνωρίζετε το πρώτο από τα δύο θέματα που έχουμε επιλέξει είναι το μέλλον της ευρωπαϊκής φορολογικής πολιτικής φορολογία, ψηφιακή οικονομία, συνέχεια των Panama Papers και των Paradise Papers και των αποτελεσμάτων της ε, Διερευνητικής Επιτροπής του Κοινοβουλίου. Όπως ξέρετε το Κοινοβούλιο ασχολήθηκε εντατικά με το θέμα αυτό και όσον αφορά την έρευνα αλλά και όσον αφορά την νομοθετική πλευρά. Ε, βεβαίως, ε, δυστυχώς, σε αυτό το τομέα ε, εμείς έχουμε απλό συμβουλευτικό ρόλο. Ο δικός σας ο ρόλος, λοιπόν, είναι ζωτική σημασίας και αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε με την νέα κοινή ενιαία φορολογική βάση και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να εξορθολογήσουμε τα ψηφιακά θέματα με την ε, ε, κοινή ενιαία φορολογική βάση των επιχειρήσεων. Ολοκληρώσαμε και την οδηγία για την ε, ε νομιμοποίηση παρανόμων εσόδων, στην οποία έχουμε συναπόφαση και θέλουμε να δούμε και τι θα γίνει με το Συμβούλιο, να περάσουμε και σε εκτενές αναχώρα. Έχουμε και το πακέτο του ΦΠΑ ε, οι ομιλητές βεβαίως ε, στο πάνελ και εσείς θα σχολιάσετε τα θέματα αυτά. Πριν ξεκινήσουμε όμως με το πάνελ θα ήθελα να δώσω το λόγο στην συμπρόεδρό μου, στον συμπρόεδρό μου, συγγνώμη, αν θέλετε να πείτε κάτι, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Γκολτιέρη. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αξιότιμοι βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων, αγαπητοί συνάδελφοι. Για μένα είναι τιμή να συμπροεδρεύω σε αυτό το πάνελ η διακοινοβουλευτική διάσκεψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση και στη διάρκεια της Βουλγαρικής Προεδρίας. Ε, ασχολούμαστε με θέματα φορολογικής πολιτικής, με ανάκτηση της εμπιστοσύνης και φορολογική δικαιοσύνη και κοινωνική δικαιοσύνη. Πρέπει λοιπόν να δούμε αποτελεσματική και δίκαιη φορολόγηση της ε, ε, ψηφιακής οικονομίας ε, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και πρέπει να δούμε και τη μεταρρύθμιση των εθνικών κανόνων για την ε, κατανομή των κερδών και άλλους κανόνες που ισχύουν για την ψηφιακή τεχνολογία. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξετάσουμε και την πρόταση για την ενιαία κοινή φορολογική βάση ε, επιχειρήσεων ε, των, ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χαιρόμαστε που θα γίνει αναθεώρηση των κανόνων της έδρας της επιχείρησης και θα δούμε και πώς μπορούμε να έχουμε ένα τύπο βάσει του οποίου θα λαμβάνουμε υπόψη πού έχουν γίνει τα κέρδη και πού βρίσκονται τα στοιχεία του ενεργητικού. η εναρμόνιση της φορολόγησης ε, θα αυξήσει την εμπιστοσύνη ε, των πολιτών ε, στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης θεωρούμε ότι πρέπει να δούμε τα θέματα νομοποίησης παρανόμων εσόδος, το ξέπλυμα και τη φοροδιαφυγή, και γιατί πρέπει να λάβουμε αποφασιστικά βήματα στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον συμπρόεδρό μου. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο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 υλοποιηθεί μέχρι τώρα σε θέματα φορολογικής πολιτικής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από την αρχή αυτής της θητείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την οποία προεδρεύει ο Πρόεδρος Γιούνκερ και καθώς επίσης να αναφερθώ στις βασικές προκλήσεις που ε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε προκειμένου να ολοκληρώσουμε την εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Πιστεύω ότι είναι χρήσιμο να ξεκινήσουμε δίνοντας έμφαση στην εξαιρετική συνεργασία που υπάρχει σε διοργανικό επίπεδο μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και με πολλά εθνικά κοινοβούλια με τα οποία είχαμε και ε, ε, καρποφόρους διαλόγους ε, που βοήθησαν στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος και είχαν και ιδιαίτερη βαρύτητα στην απόφαση που λαμβάνουν τα Συμβούλια Υπουργών σε θέματα φορολογίας, διότι όπως υπενθύμησε ο πρόεδρος Γκουαλτιέρη, η νομοθετική διαδικασία στον τομέα της φορολογίας απαιτεί ομοφωνία στο Συμβούλιο. Το πρώτο στοιχείο που είναι αρκετά αξιοσημείωτο είναι το θέμα της φορολογικής διαφάνειας. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι από την αρχή αυτής της θητείας τα όσα καταφέραμε όσον αφορά την έγκριση νομοθετικών κειμένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να βελτιώσουμε τη φορολογική διαφάνεια, είτε πρόκειται στον τομέα της ανταλλαγής ε, των tax rulings, είτε πρόκειται ε, στη, για τις εκθέσεις αναχώρα για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Οι πρόοδοι που έχουν επιτευχθεί στα πλαίσια της οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων και το τέλος του τραπεζικού απερίτου μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών τραπεζικού χαρακτήρα ε, αποτελούν νομοθετικά κείμενα τα οποία θα επιτρέψουν στις φορολογικές ε, αρχές ε, να διαθέτουν πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες ε, προκειμένου να γίνεται σωστά η συλλογή των φόρων. Ε, εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαγρυπνά, διότι θα πρέπει να επαληθεύσουμε ότι θα γίνει σωστή μεταφορά και εφαρμογή από τα κράτη-μέλη, διότι ο στόχος μας ε, βεβαίως ε, δεν είναι απλώς να εγκρίνονται κείμενα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να εξασφαλίσουμε ότι εφαρμόζονται σωστά αυτά τα κείμενα σε επίπεδο χωρών. Ο δεύτερος τομέας στον οποίο έγιναν σημαντικές πρόοδοι είναι η ενίσχυση της νομοθεσίας που επιτρέπει την καταπολέμηση ε, της φοροδιαφυγής ε, και της επιθετικής φορολογικής πρακτικής. Ε, είχαμε δύο οδηγίες εδώ, οι οποίες είναι στη διαδικασία μεταφοράς από πλευράς κρατών μελών, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις επιχειρήσεις που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν κάποιες φορολογικές ευκαιρίες για να αποφύγουν την καταβολή των φόρων και να μειώσουν την ε, νόμιμη φορολογική βάση των ε, κρατών μελών μας. Ο τρίτος τομέας είναι το εξωτερικό σκέλος ε, αυτού του θεματολογίου, διότι θεωρήσαμε ότι ήταν χρήσιμο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσουμε να εμπλουτίσουμε αυτό το θεματολόγιο για τη διαφάνεια και την χρηστή φορολογική διαχείριση και σε εξωτερικό επίπεδο, πέραν των συνόρων μας. Γι' αυτό ακριβώς και ε, κάναμε πολλά ώστε το Συμβούλιο να εγκρίνει, όπως και έκανε τον Δεκέμβριο, ένα κατάλογο ε, με ε, φορολογικές επικράτειες οι οποίες δεν είναι συνεργάσιμες, ώστε να μπορέσουμε να ασκήσουμε και πίεση ε, σε αυτές τις φορολογικές επικράτειες οι οποίες δεν τηρούν τα βασικά πρότυπα και προδιαγραφές που έχουν συμφωνηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο αποτέλεσμα αυτής της διαδικασία είναι κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό, διότι ε, ως αποτέλεσμα αυτών των εργασιών, πέραν αυτής της μαύρης λίστας ε, με τις φορολογικέ επικράτειες που δεν συνεργάζονται, υπάρχουν 55 ε, ε, φορολογικές επικράτειες, τρίτες φορολογικές επικράτειες που δεσμεύτηκαν να επανεξετάσουν το νομοθετικό και κανονιστικό τους πλαίσιο ώστε να συμμορφωθούν προς τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από την υλοποίηση αυτών των δεσμεύσεων είχαμε περίπου 600 νέες συμφωνίες ε, ανταλλαγής πληροφοριών και 100 φορολογικά καθεστώτα τα οποία είναι υπό εξέταση και αυτά θεωρούμε ότι αποτελούν πρόοδο. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τις πρόοδους μας εν γέννη. Για το μέλλον έχουμε δύο μεγάλα προγράμματα στα σκαριά. Το πρώτο είναι η έγκριση της ε, κοινή ε, φορολογικής βάσης των επιχειρήσεων, κάτι το οποίο αποτελεί και... Ε, ένα από τα θέματα τα οποία απασχολεί το Κοινοβούλιο ε, και φυσικά η ψηφιακή οικονομία, διότι πλέον πρέπει να δούμε τις νέες μορφές επιχειρήσεων για να μπορέσουν να δημιουργήσουν ε, κέρδη και αξία και να βρίσκονται στην εσωτερική αγορά με φορολογικές βάσεις οι οποίες θα ανταποκρίνονται καλύτερα στα όσα κάνουν οι επιχειρήσεις. Αυτά είναι τα δύο έργα που έχουμε στα σκαριά που με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων που αντιμετωπίζουν τις ίδιες προσδοκίες από πλευράς πολιτών σε επίπεδο χώρας. Ε, προσπαθούμε να έχουμε κάποια αποτελέσματα μέχρι το τέλος της θητείας και ε, τη λήξη της εντολής της παρούσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βέρνερ Λάγκε, πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για τα έγγραφα του Παναμά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ εν συντομία στα πορίσματα της Εξεταστικής Επιτροπής ε, Πάνα, των εγγράφων του Παναμά, έπειτα από τις δημοσιεύσεις που έγιναν από το Wikileaks το 2010, Offshore Leaks 2013, Lux Leaks 2014, Swiss, Leaks 2016, ε, τον Απρίλιο, του 15, τον Απρίλιο του 2016 ε, δημοσιεύθηκαν 2,6 τεραμπάιτ εγγράφων από δικηγορική εταιρεία που είχε την έδρα της στον Παναμά και περιείχε πολλές πληροφορίες σχετικά με 120.000 ε, εταιρείες ταχυδρομικές θηρίδες ήταν μια τεράστια διαρροή εμπιστευτικών δεδομένων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπειτα από δύο εξεταστικές επιτροπές, τάξε 1 και τάξε 2, αποφάσισε να συστήσει εξεταστική επιτροπή στις 8 Ιουνίου του 2016 και ε, καθώς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, οι εξεταστικές επιτροπές έχουν διάρκεια το ανώτατο 18 μήνες τον Δεκέμβριο του 2017 οι εργασίες της Επιτροπής ολοκληρώθηκαν. Στη διάρκεια αυτή διοργανώσαμε 26 ακροάσεις, αναθέσαμε την εκπόνηση μελετών και πραγματοποιήσαμε 8 συνολικά αποστελές. Τη ΣΥΠΑ, τη Μάλτα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πορτογαλία, την Ελβετία, την Κύπρο και στο τέλος άλλη μία φορά στη Μάλτα στη βάση των αποφάσεων του Κοινοβουλίου σχετικά με την τήρηση των αρχών του κράτους δικαίου στη χώρα αυτή. Ακούσαμε πολλές φορές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τρεις φορές ήρθε ο κύριος Μοσκοβισή στην Εξεταστική Επιτροπή, δύο φορές η Επίτροπος Επίτροπος και μία φορά μάλιστα ήρθε και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Γιούγκερ και θεωρώ ότι αν έχει κανείς ε, παρακολουθήσει τις φορολογικές εξελίξεις τα τελευταία χρόνια τότε σίγουρα θα έχει διαπιστώσει και την ε, δραστηριοποίηση στον τομέα αυτό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάτι που έχει οδηγήσει και σε μια συνολική ε, αλλαγή στη στάση διαφόρων πλευρών. Αυτό που μέχρι, τότε, μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν ως επιχειρηματικό μοντέλο που αφορά την, κάθε χώρα ξεχωριστά και εκεί που δεν δεν συζητιόνταν καθόλου τα ζητήματα της κατανομής ε, ή των φορολογικών βαρών ή της δικαιοσύνης των φορολογικών συστημάτων ή και της δίκαιης κατανομής ή του επιμερισμού των φορολογικών βαρών ε, και εκεί που θεωρούνταν πριν, μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεμητό να προσπαθεί κάθε χώρα να ε, δημιουργεί φορολογικά ωφέλη για τον εαυτό της. Ε, χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι το Λουξεμβούργο το οποίο για, δεκάδ για δεκαετίες αποτέλεσε τον κορβανά στον οποίο κατέληγαν μαύρα χρήματα μεγάλων επιχειρηματών πολιτικών ομήλων από τις δραστηριότητές τους σε ολόκληρο τον κόσμο. Εμείς λοιπόν καταφέραμε μέσα από τη συζήτηση που ξεκινήσαμε με δική μας πρωτοβουλία να υπάρξει μια αλλαγή νοοτροπίας, κάτι που επηρέασε και συγκεκριμένα άτοπα και ε, καταφέραμε με αυτόν τον τρόπο να ε, σπάσουμε αυτόν τον φαύλο κύκλο της ε, διαρκούς και αέναης μεταμόρφωσης των φορολογικών προσώπων και ταυτοτήτων διαφόρων εταιριών. θέσαμε λοιπόν κέρια ερωτήματα τα οποία αφορούσαν τη συμπεριφορά των κρατών μελών αλλά όχι μόνο. Στα δεδομένα μάλιστα που ζητήσαμε είχαμε κράτη-μέλη τα οποία προσπάθησαν να μπλοκάρουν το δρόμο μας. Είχαμε την ομάδα Code of Conduct για παράδειγμα που είναι μια διακυβερνητική επιτροπή των κρατών μελών και όχι ευρωπαϊκός θεσμός η οποία μάλιστα αρνήθηκε να προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή ακριβώς με την αιτιολόγηση ότι δεν είναι ευρωπαϊκός θεσμικό, θεσμικό όργανο με επικεφαλής μάλιστα μια ε, Ιταλίδα τεχνοκράτησα. Μας δόθηκαν κάποια στοιχεία με διαγραμμένα όμως τα σημαντικότερα και πιο κρίσιμα σημεία. Ε, κάποιες φορές μάλιστα λαμβάναμε ε, έγγραφα που, περιλάμβαναν μόνο την ημερήσια διάταξη χωρίς καμία, ε, κανένα ουσιαστικό περιεχόμενο στα οποία συνέρχονταν και συνεδρίαζαν στο πλαίσιο της Επιτροπής αυτής τα κράτη-μέλη, χωρίς βεβαίως συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και εκεί φαίνεται ότι υπήρχαν συζητήσεις για συγκεκριμένε, χώρες, ακόμα και συγκεκριμένε περιφέρειες συγκεκριμένων χωρών, όπως στην περίπτωση της Ισπανίας για παράδειγμα, ε, κάτι που βεβαίως πρέπει να σας πω ότι μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι δυστυχώς οι εργασίες μας δεν στέφτηκαν με την επιτυχία που θα μπορούσαν να είχαν ε, αν είχαμε τη συνεργασία όλων των φορέων και όλων των ε, πλευρών που είχαμε προσκαλέσει. Να σας ε, ενημερώσω ότι υπήρξαν, είχαμε συνολικά εννέα αρνήσεις ε, προσέλευσης. Αυτό βεβαίως πρέπει να αλλάξει με την επόμενη τροποποίηση της συνθήκης. Ο πρόεδρος τόνισε ήδη ότι υπάρχουν ήδη στην πορεία ε, μια σειρά από νομοθετικές προτάσεις ε, οι οποίες, ε, στις οποίες έχουν ληφθεί υπόψη τα πορίσματα της Εξεταστικής μας Επιτροπής για παράδειγμα η κοινή φορολογική βάση εταιριών οι συστάσεις αναχώρες οι κανόνες διαφάνειας για τον φορολογικό σχεδιασμό, οι πληροφοριοδότες, ευρωπαϊκός κατάλογος των μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών και σε αυτό το τομέα είχαμε ένα πρόβλημα ως Εξεταστική Επιτροπή με το Συμβούλιο ε, ε, Υπουργών Οικονομίας που ε, κατάρτισε αυτόν τον κατάλογο για τρίτες χώρες όμως αρνήθηκε να εντάξει τα τέσσερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα έπρεπε να βρίσκονται σε αυτόν τον, κατάλογο και είναι οι τέσσερις εξής χώρες. Η Ιρλανδία λόγω των ειδικών ρυθμίσεων βλέπε Apple ε, ε, κάτω χώρες λόγω των ε, αδειών χρήσης που εκδίδει, Λουξεμβούργο λόγω των tax rulings και Μάλτα λόγω του συνολικού φορολογικού συστήματος της χώρας αυτής και εδώ νομίζω ότι το πρώτο θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει είναι η διαφάνεια, δεύτερον η συνεργασία μεταξύ των φορολογικών αρχών, τρίτον η υλοποίηση και η εφαρμογή των διεθνών κανόνων, τέταρτον ε, το ερώτημα πώς στο μέλλον και εδώ δεν μιλάμε για, εθνική κυριαρχία, πώς στο μέλλον θα ε, φορολογούνται τα κέρδη των ε, γιγάντων του διαδικτύου. Η Apple και μόνο έχει ε, ε, κρύψει 4,5 δισεκατομμύρια κέρδη σε φορολογικούς παραδείσους. Πώς λοιπόν θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τη φορολόγηση αυτών των κερδών από τα κράτη-μέλη. Είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολήσει και τα εθνικά κοινοβούλια και τα απασχολεί ήδη. Άλλωστε είναι ένα θέμα μεταξύ άλλων και αναπτυξιακής πολιτικής. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από την Αφρική να κάνει βήματα Βελτίωση βελτίωση στον ε, τομέα ε, τη διακυβέρνηση, για παράδειγμα όταν εμεί οι ίδιοι δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε τις μεγάλες, τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και τις πολυεθνικές να καταβάλουν του φόρου ε, τους φόρους τους στις αφρικανικές χώρες. Σταματώ εδώ και θα έχουμε βεβαίω ευκαιρία να συζητήσουμε περαιτέρω αυτό το θέμα. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Δυστυχώς βρισκόμαστε υπό χρονικό περιορισμό. Έχουμε και, άλλο θέμα να συζητήσουμε. Έχουμε και το δείπνο στις 7. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Έρικ Φούρτερ που είναι ε, ε, πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της ε, Γαλλικής Εθνοθυνέλευσης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα επικεντρωθώ στην ψηφιακή οικονομία. Η ΚΑΦΑ είναι σήμερα εξίσου δυνατές όπως και οι χώρες μέλη. Και οι χώρες μάλλον, όπως και τα κράτη. Υπάρχει σε αυτές μια οικονομική δυνατότητα που ξεπερνάει εκείνη κρατών και έχουν και την δυνατότητα να συλλέγουν στοιχεία, δεδομένα με μοναδικό τρόπο σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε σήμερα που βρίσκεται μέσα σε συνεχείς αλλαγές. Στη Γαλλία λοιπόν προσέχουμε πάρα πολύ τα θέματα της, ε, των αδικιών. Αδικιών μεταξύ των χωρών για να επανέλθω σε κάτι που είχε πει ο Λέα Λαμασούρ στην ε, δικιά μας ε, εθνοσυνέλευση πριν από λίγο καιρό, ήταν τελικά ποιος είναι που κλέβει, γιατί δεν πρόκειται μόνο για το κοινωνικό dumping. υπάρχουν πολύ περισσότερα πράγματα. Φυσικά και υπάρχουν σκάνδαλα, Wikileaks, ε, Panama Papers, εξού και εξεταστική επιτροπή, στην οποία αναφέρθηκε ο συνάδελφος, εγώ θα έλεγα ότι είναι κρίμα που τελικά είναι οι δημοσιογράφοι που μας οδηγούν να κάνουμε αυτές τις έρευνες. Θα έπρεπε στα, σε εθνικό επίπεδο να ανεβάσουμε ταχύτητα. Έχω σήμερα λοιπόν την αίσθηση ότι ε, περιορίζομαι από διάφορες επιχειρήσεις. Όταν το Facebook με 30 εκατομμύρια ε, στη Γαλλία πληρώνει τόσο λίγους φόρους, υπάρχει ζήτημα. Όταν το Google με διοικητικές αποφάσεις δεν αναγκάζεται να πληρώνει το ίδιο. Το ίδιο και για την Amazon και για άλλους. Οπότε οι ευρωπαϊκοί κανόνες, πρώτα απ' όλα οι εθνικοί κανόνες των χωρών, αλλά και στη συνέχεια οι ευρωπαϊκοί κανόνες, θα συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή, και γενικότερα οι κανόνες του ΩΣΑ, γιατί εγώ πιστεύω στον ΩΣΑ, εδώ έχουμε να κάνουμε παγκόσμιες επιχειρήσεις, άρα λειτουργούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι κανόνες που διέπουν την λειτουργία τους θα πρέπει να είναι κάτι το σωστό. Μια επιχείρηση σήμερα, όπως και αν παράγει όποιο σύστημα παραγωγής και αν έχει, θα πρέπει να υποβάλλεται σε φορολογία με τον ίδιο τρόπο όπως και άλλες. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, το ακούσαμε και πριν. Η Γαλλία έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαφάνεια. Πριν από καμιά δεκαριά χρόνια, ...όσα με την Ευρώπη δεσμεύτηκαν στην καταπολέμηση της απάτης σε διεθνές επίπεδο. Πώς να έχουμε λοιπόν αυτή την φορολογική δικαιοσύνη, πώς να τη ρυθμίσουμε. Έχουμε μια έκθεση που ετοίμασα με συναδέρφους πριν από λίγο καιρό στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση και λέμε ότι πρέπει να ξαναβάλουμε τις βάσεις που λένε ότι εκεί που υπάρχουν τα κέρδη, εκεί πρέπει και να πληρώνονται οι φόροι. Η δουλειά που γίνεται σήμερα για το είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί προβλέπει την εναρμόνιση στον υπολογισμό των κερδών. Πρέπει όμως επίσης να πάμε και πολύ γρήγορα. Πρέπει να διευκρινίσουμε τι είναι κάποια ευρυδικά προϊόντα να διευκρινίσουμε και να κάνουμε πιο αυστηρούς τους κανόνες της μεταφοράς των κερδών και επίσης χρειαζόμαστε και φορολογική σταθερότητα. Η Γαλλία το χρειάζεται, μπορεί να μην ισχύει απαραίτητα στις χώρες σας, αλλά η Γαλλία το χρειάζεται, γιατί στη Γαλλία αλλάζουν συχνά οι κανόνες. Όμως σε αυτό το τομέα δεν πρέπει να υπάρχει ακινησία γιατί η δυνατότητα φορολόγησης είναι πολύ πιο αργή σήμερα από ό,τι η εξέλιξη των οικονομιών. Οι φορολογικοί κανόνες δηλαδή εξελίσσονται πιο αργά από ό,τι η ίδια οικονομία. Άρα πρέπει να επιλέξουμε κάποιες βάσεις και φυσικά μπορούμε να συζητήσουμε για πολύ, αλλά η Γαλλία έκανε προτάσεις όπως και άλλες χώρες με διάφορες ιδέες, φορολόγηση, βάση του τζίρου. Εντάξει, είναι συζητήσιμο. Να το συζητήσουμε. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια μειονεκτήματα σε αυτό, αλλά δεν λέω ότι θα είναι και ο τελικός ο στόχος. Πάντως, αν μη τι άλλο έχει κάποιο ενδιαφέρον να συζητηθεί, γιατί μπορεί βραχυπρόθεσμα να είναι μια λύση, πριν συζητήσουμε μια άλλη λύση πιο μακροπρόθεσμη. Πάντως, οι ψηφιακές επιχειρήσεις σήμερα αποτελούν μονοπόλια. Συγκεντρώνουν κέρδη χωρίς να πληρώνουν φόρους και από τα κέρδη αυτά πηγαίνουν και αγοράζουν άλλες επιχειρήσεις σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Ε, δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε αυτό το πράγμα να συνεχιστεί. Άρα χρειαζόμαστε πρώτα μια λύση βραχυπρόθεσμη και αν είναι ολοκληρωμένη, έχει καλό Αν δεν υπάρχει τέτοια ολοκληρωμένη λύση, α έχουμε μια διάμεση λύση. Για να μπορέσουμε να φορολογήσουμε τα κέρδη. Και υπάρχουν και άλλου είδους επιχειρήσεις εκτός από τις γκαφά. Τα Airbnb για παράδειγμα. Και είναι και αυτή μια κατηγορία επιχειρήσεων σχετικά με την οποία πρέπει να γίνουν και άλλες προτάσεις στη Γαλλία, κάναμε κάποιες ώστε όποιος νοικιάζει το διαμέρισμά του και ε, με το Airbnb και αυτός που το νοικιάζει με πιο παραδοσιακό τρόπο να φορολογούνται εξίσου με τον ίδιο τρόπο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο Μέντλα έχει τώρα το λόγο, ο οποίος είναι πρόεδρος της Επιτροπής Panama Papers στο Βελγικό Κοινοβούλιο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που ασχολείστε με τα Panama Papers και τις εργασίες ε, της Επιτροπής ε, ε, στην οποία είχα την τιμή να προεδρεύσω στο Βελγικό Κοινοβούλιο. Να πω δύο λόγια για τις ψηφιακές επιχειρήσεις. Το πρόβλημα είναι αρκετά σημαντικό. Το Amazon και το Alibaba, για να αναφερθώ σε δύο, έχουν ένα τζίρο εργασίας ο οποίος είναι ισοδύναμος με το ΕΠ του Βελγίου. 450 δις δολάρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε ε, σημαντικές προκλήσεις. Το θέμα είναι ότι αν δεν είμαστε σε θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο να έχουμε μια βάση κεφαλαιοποίηση, θα πρέπει κατά την άποψή μου να δούμε τον κύκλο εργασιών. Ε, δεν θεωρώ ότι υπάρχει άλλη λύση βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα να προσπαθήσουμε να δούμε τις ροές των χρημάτων, δηλαδή τον κύκλο εργασιών στις χώρες προορισμού των αγαθών ή των υπηρεσιών που παρέχονται. Και βεβαίως ε, ε, λαμβάνοντας υπόψη και τη δυνατότητα ενίσχυσης της ε, φορολογικής εναρμόνισης ε, για να μπορέσουμε να δούμε πού βρίσκονται τα κύρια κέρδη των επιχειρήσεων. Ξέρουμε ότι είναι βέβαια πολύ δύσκολο αυτό. Όσον αφορά τα Panama Papers, όντως το Βελγικό Κοινοβούλιο ασχολήθηκε με το θέμα σχετικά γρήγορα και το πρώτο ε, όφελος που προέκυψε από αυτό είναι ότι οι βουλευτές ε, που ε, ζήτησαν από το Κοινοβούλιο να συζητήσει το θέμα, επέτρεψαν στην πραγματικότητα να επιταχύνουμε τα θέματα για τους φορολογικούς παραδόσους, για να δούμε και την φοροδιαφυγή, αλλά και πλέον η εκτελεστική εξησία ξεκίνησε 200 ε, υποθέσεις όσον αφορά ε, τα θέματα που απασχολούν το Βέλγιο όσον αφορά το σκάνδαλο των Panama Papers και η δικαιοσύνη από πλευρά τη, ε, ο εισαγγελέα πιο συγκεκριμένα, ξεκίνησε πάνω από 300 υποθέσεις. και είναι 200 στο Κοινοβούλιο και 300 γιατί μπορεί πολλαπλές περιπτώσεις να αφορούν τις ίδιες επιχειρήσεις ή το δικαιούχο. μεταξύ 200 δηλαδή και 300 υποθέσεων αν άνοιξαν και εξετάζονται από τι διάφορε υπηρεσίε του κράτου. Δεν αρκούσε βέβαια αυτό, έπρεπε το Κοινοβούλιο να κάνει και έναν απολογισμό για το συσχετισμό των δυνάμεων και τι δυνατότητε έχουμε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των φορολογικών παραδείσων. Και ακριβώ για αυτό το λόγο έγιναν αρκετέ ακροάσει, ε, περίπου 90 ώρε ακροάσεων, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ε, πέραν των ομάδων εργασία που είχαμε για να δούνε τι διάφορε εκθέσει, να εξετάσουν τα θέματα και Ακούσαμε όλες τις υπηρεσίε του κράτους, ε, τις φορολογικές αρχές, τον εισαγγελέα βεβαίως, τις αστυνομικές αρχές, αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω του κυρίου Λάγκεν, ο οποίο ήταν αρμόδιο για τι εργασίε τη Επιτροπή Πάνα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επίση τον Αντιπρόεδρο του Παναμά, ο οποίο ήταν σε επίσημη επίσκεψη εδώ στο Βέλγιο και μα έκανε την τιμή να έρθει να απαντήσει σε ερωτήσει μα. Και επίσης ε, ε, και αρκετού οργανισμού και ιδρύματα, και αυτό είναι σημαντικό, που με τον, ένα, με τον άλλο τρόπο ασχολούνται με τον έλεγχο του χρηματοπιστωτικού τομέα. Ε, η Εθνική Τράπεζα φυσικά, γιατί αυτό είναι ο ρυθμιστή και ο επόπτης ε, των τραπεζών και είναι πολύ σημαντικό και όπως ξέρετε είναι πολύ δύσκολο να ε, υπάρχει ένας κύκλος απάτης αν δεν υπάρχει ένας χρηματοπιστωτικός κύκλος. Επομένως πρέπει να δούμε το χρηματοπιστωτικό κύκλο, δηλαδή τις τράπεζες, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αλλά φυσικά και τις διαδικασίες ξεπλήματος. Από εκεί προέκυψαν μια σειρά από συστάσεις, οι οποίες ε, δεν έτυχαν βέβαια γενικότερη πολιτική συνένεση, διότι αυτομάτως βεβαίως γνωρίζετε το θέμα της ε, φορολογίας, είναι δείγμα των διαφωνιών που υπάρχουν σε πολιτικό επίπεδο αλλά παρόλα αυτά μπορούμε να πούμε ότι έχει υπάρξει κάποια πρόοδος ω προ την ανάγκη να υπάρχει ένα καθεστώς, ε, να υπάρχει ένα εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματο. Αυτή είναι μια διαφορά που έχουμε σε σχέση ε, με τη Γαλλία. Δεν έχουμε εισαγγελέα αρμόδιο μόνο για χρηματοπιστωτικά ζητήματα. Θα έπρεπε να έχουμε έναν ε, ειδικό στον οποίο θα μπορούσαμε να αποτανθούμε όταν πρόκειται για ένα τέτοιο θέμα. Υπάρχει όμως μια αξιοσημείωτη πολιτική συνένεση για να υπάρχει ένας πραγματικός εισαγγελέα ε, χρηματοπιστωτικών οικονομικού εγκλήματος ε, που να ασχολείται μόνο ε, για, σε θέματα αυτά φοροδιαφυγής πιο συγκεκριμένα και φορολογικής απάτης. Και φυσικά υπάρχουν και διάφορες υπηρεσίες και εδώ επειδή υπάρχει διαφωνία δεν υπάρχει συμφωνία προς τα μέσα που θα πρέπει να δώσουμε στις διάφορες υπηρεσίες. Υπάρχει και συνένεση όμως για την ανάγκη να επιταχύνουμε την εφαρμογή των ε, ε, ευρωπαϊκών ε, νομοθετημάτων που επιτρέπουν την διαδικασία αυτή, κυρίως το θέμα του πραγματικού δικαιούχου, ένα θέμα που ίσως γνωρίζετε καλά και φυσικά ιδιαίτερα προσοχή όσον αφορά την ε, δυνατότητα ε, διεύρυνσης ε, των αρμοδιοτήτων μας. Δεν ασχοληθήκαμε με το transfer pricing, την τιμή μεταβίβασης, το ελέγξαμε ακροθυγώς. Πιστεύουμε ότι θα μπορούσαμε να διευρύνουμε τις προθεσμίες φορολόγησης που έχουν στη διάθεσή τους οι φορολογικές αρχές για να καταπολεμήσουμε τη συγκεκριμένη μορφή φορολογικής απάτης. Ε, θέλουμε να το διευρύνουμε στα 10 χρόνια αντί τα 7 που έχουμε αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιες συναλλαγές οι οποίες περνούν μέσα από ένα φορολογικό παράδεισο. Αυτά κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο. Υπάρχουν λοιπόν ε, ε, πράγματα αρκετά να κάνουμε, υπάρχουν κάποιες συστάσεις τις οποίες απευθύναμε προς το Κοινοβούλιο, για να, το κυβέρνηση για να καταρτήσει έναν οδικό χάρτη και εμείς ως βουλευτές θα πρέπει να ελέγξουμε ότι όντω η εκτελεστική εξουσία θα υλοποιήσει όλες αυτές τις ε, προτάσεις. Ευχαριστούμε πολύ τους ομιλητές. Το λόγο έχει ο κύριος Κάνεφ και πρέπει να σας πω ότι το επόμενο θέμα θα αρχίσουμε να το συζητάμε στις 6, οπότε σας παρακαλώ να είστε πάρα πολύ σύντομοι. Δεν είμαι βέβαιος αν θα καταφέρουμε να δώσουμε το λόγο σε όσους τον έχουν ζητήσει. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Ε, ναι, Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να περιοριστείτε όλοι στα δύο λεπτά. Ο κύριος Σταϊκούρας έχει το λόγο για δύο λεπτά. Πρώτος ομιλητής. Κάθε φορολογικό σύστημα πρέπει να διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας, της ουδετερότητας, της απλότητας, της σταθερότητας, της λειτουργικότητας, της ισορροπίας, της ισότητας και να στοχεύει στην οικονομική ανάπτυξη. Δυστυχώ, διαχρονικά και διατοπικά εμφανίζονται εμπόδια στην επίτευξη αυτών των στόχων, ενώ οι νέε τεχνολογίε και η αλματώδη αύξηση των συναλλαγών μέσω ψηφιακών πλατφορμών αυξάνουν τι προκλήσει για τη φορολογική διοίκηση. Για την αντιμετώπιση αυτών απαιτείται η υλοποίηση ενό συνεκτικού πλέγματο πολιτικών, όπω είναι ενδεικτικά τέσσερι άξονε. Ο πρώτο είναι η εφαρμογή ενό ενιαίου με απλούστορους κανόνες και χαμηλότερους συντελεστές ευρωπαϊκού χώρου ΦΠΑ που θα παρέχει ευελιξία και θα δημιουργεί ένα καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ο δεύτερος είναι η ενίσχυση της συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών και η εναρμόνιση των πλαισίων φορολογίας με κοινή φορολογική βάση, όπως είπατε, για τις επιχειρήσεις, ώστε να εξασφαλιστεί ισόρροπη ανάπτυξη και ευημερία. Τρίτο άξονα είναι η δημιουργία ενό πιο αυστηρού και αποτελεσματικού πλαισίου αντιμετώπιση καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών μέσω των φορολογικών παραδείσων, με τη συμμετοχή στα δίκτυα που έχουν δημιουργηθεί και τι ομάδε εργασία για να αντιμετωπιστούν φαινόμενα τύπου Panama Papers, εξετάζοντα θέματα που σχετίζονται με τον πραγματικό δικαιούχο, την φορολογική κατοικία και το διακριτικό προφίλ των φορολογουμένων. Και τέλος, τέταρτον, η εναρμόνιση των κανόνων πράγματι σε παγκόσμιο επίπεδο για την ψηφιακή οικονομία, ώστε το κέρδος, όπως σωστά αναφέρατε, να φορολογείται στον τόπο στον οποίο παράγεται. Αρχικά με την προσωρινή λύση της επιβολής φόρου διαδικτύου επί του κύκλου εργασιών αυτών των εταιριών και στη συνέχεια εναρμονίζοντας τις νομοθεσίες των κρατών με το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, κάνοντας πιο αυστηρούς τους ελέγχους για τη μεταφορά κερδών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκάλι από την Ιταλία έχει το λόγο. Thank you, Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι έχουμε προβλήματα πολλά. Αλλά δεν πρέπει να υποτιμούμε και την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε επίπεδο ΩΣΑ αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να αναφερθώ σε τρία σημεία. Συστάσεις και εκθέσει αναχώρα που έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο ΩΣΑ. Αυτόματη ενταλλαγή πληροφοριών. Πρόκειται για επανάσταση όσον αφορά την ε, συλλογή φόρων. Έμεση φορολογία Τρίτο στοιχείο. Έχουμε συμφωνήσει σε επίπεδο ΩΣΑ επί των αρχών της χώρας προορισμού, εκεί όπου γίνεται η κατανάλωση, εκεί πληρώνεις τον έμεσο φόρο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι το 20 ή το 22% των πωλήσεων είναι σημαντικότερο από τους φόρους επί των κερδών. Όχι ότι δεν πρέπει βεβαίως να συλλέγονται και αυτοί. Να σας πω κάτι ακόμη, γιατί στο Ιταλικό Κοινοβούλιο έχουμε συζητήσει πολύ και έχουμε καταλήξει σε μια απόφαση. Ό,τι και αν κάνεις, νομίζω ότι ο Βέλγος συνάδελφος μόλις το είπε, είναι πολύ σημαντικό. Στο τέλος πρέπει να καταλήγεις σε φόρο επί των πωλήσεων. Κάτι που είναι πολύ παρόμοιο με έμεσο φόρο και ο ΩΣΑ στα μέσα Μαρτίου θα ε, υποβάλει και τις δικές του συστάσεις, προτάσεις για κάθε χώρα συγκεκριμένα και θα δείτε εκεί ότι η μόνη βιώσιμη λύση είναι η φορολόγηση των πωλήσεων. Υπάρχουν δύο προβλήματα βεβαίως. Πρώτον, ότι όπως και στους ε, έμεσους φόρους οι καταναλωτές θα είναι εκείνοι που θα κληθούν να καταβάλουν τους φόρους αυτού και όχι οι μεγάλες ε, εταιρείες του διαδικτύου και δεύτερον καταλήγεις να φορολογείς την καινοτομία. Όλες οι χώρες μας προσπαθούν να δώσουν κίνητρα στην ψηφιακή καινοτομία και ταυτόχρονα ε, καταλήγουμε να την πληρώνουμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεφύγει κανείς από αυτήν την παγίδα που μόλις περιέγραψα. Ευχαριστώ πολύ και που τήρησατε το χρόνο. Ο κύριος Βαλαούρας από την Ελλάδα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην Ελλάδα έχουμε μία παροιμία που λέει τον ξέρουμε τον ένοχο και είναι γνωστή αιτία. Και στην προκειμένη περίπτωση μια και συζητούμε για την απόκρυψη τεράστιων κερδών και για από την ψηφιακή οικονομία Αναφέρθηκε ήδη η ομάδα Κόντακ που αντιδρά στην εξυγίανση. Ε, εννιά κράτη έχουν αρνηθεί να προσέρθουν καν στην Εξεταστική Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου και τέσσερα τουλάχιστον κράτη όπως η Ινλανδία, Ολλανδία, Λουξεμβούργο και Μάλτα δεν ε, συνεργάζονται για διαφάνεια, για γενικότερη συνεργασία, κοινοποίηση στοιχείων κτλ. Ουσιαστικά οδηγούν σε μια πλεονεκτική θέση τις χώρες τους και κάνουν κοινωνικό ντάμπινγκ. Η ΑΠ 4,5 δις έχει κρύψει από τα κέρδη της. Και η Amazon μαζί με την Αλή Μπαμπά έχουν κέρδη όσο το ΑΕΠ του Βελγίου. Τεράστια πράγματα. Και εμείς κάνουμε συστάσεις πώς θα πρέπει οι χώρες της ε, Αφρικής να λειτουργούν. Πρόσφατα στην Ελλάδα συζητάμε το σκάνδαλο Νοβάλτης, όπου επηρεάσανε τις τιμές η χώρα μας, όχι μόνο στην Ελλάδα αυτή καθεαυτή, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε 50 άλλα κράτη παγκοσμίω. Με ένα πλέγμα διαφθοράς πολιτικών, δημοσίων υπαλλήλων, γιατρών και όπως υπόθηκε και πρέπει να μπει μια τάξη αυτά, υπάρχει, μια, υπάρχει παραγραφή πολλών αδικημάτων προχωράω και τελειώνω η ελληνική κυβέρνηση προσυπόγραψε κοινή δήλωση των υπουργών οικονομικών μαζί με 9 υπουργού που υποστηρίζουν την επιβολή φόρου άμεσα ως προσωρινή λύση τουλάχιστον για την επί του κύκλου εργασιών των εταιριών που προορισμού. Εναρμόνιση λοιπόν θέλουμε εναρμόνιση κανόνων φορολόγησης ψηφιακής οικονομίας που σήμερα κράτη έχουν διαφορετική μεταχείριση. Προτείνουμε ω πρώτο, πρώτο βήμα την παροχή πληροφοριών η κυρία Γκόμες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και μετά θα είναι Μαλτά. Γιατί αρνούνται να έχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες μέλη μία μονάδα που θα κάνει τέτοιες έρευνες. Γιατί, Γιατί πράγματι θέλουν να κρατήσουν την κατάσταση ως έχει. Ως έχει δεν πρόκειται μόνο για τη φορολογική αδικία, δεν πρόκειται μόνο για το ότι δεν έχουμε την δικαιοσύνη ή γίνεται dumping. Στην πραγματικότητα η φορολογική παράδεση που υπάρχουν και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και έξω, έτσι συνεχίζουν να μπορούν να νομοποιούν παράνομο χρήμα. Η Επιτροπή δύο χρόνια περιμένει με προτάσεις για το ΦΠΑ και μόνο έτσι θα μπορούσαμε να αποφύγουμε χρήματα να καταλήγουν στο ISIS. Αλλά τίποτα δεν γίνεται. Εγώ λέω και λυπάμαι. Εντάξει, ο ΣΑ μπορεί να είναι ένας πολύ ωραίος κόσμος, αλλά δεν κάνει τίποτα δεσμευτικό. Εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δράσουμε και οι ευρωβουλευτές μαζί με τους εθνικούς βουλευτές έχουμε τεράστια ευθύνη για να προστατεύσουμε τους πολίτες που μας εξέλεξαν και πρέπει να καταργήσουμε αυτούς τους φορολογικούς παραδείσους. Πρέπει να κάνουμε όλα αυτά που αναφέρθηκαν, που τα γνωρίζουμε καλά, ε, τα Μητρώα, την ε, καταγραφή των επιχειρήσεων, την ε, κοινή φορολογική βάση κλπ. κλπ. Πάρα πολύ ωραία πράγματα στην νομοθεσία, αλλά τίποτα δεν εφαρμόζεται. Πρέπει οι φορολογικές διοικήσεις να έχουν τους πόρους που χρειάζονται για να κάνουν ελέγχους. Να υπάρξει επίσης φορολόγηση στις τραπεζικές συναλλαγές. Και όσε δεν φτάνει. Και όλα αυτά πρέπει να γίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει την αρχή γιατί θα κάνει τη διαφορά. Κλείνει το μικρόφωνο της ομιλήτριας, την διακόπτη ο Πρόεδρος. Ξεπεράσατε το χρόνο σας. Μάλτα τώρα. Και μετά Γαλλία Γκάμπλετς. Παρακαλώ. Μάλτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα αρχίσω επαναλαμβάνοντας πρώτα απ' όλα την τοποθέτησή μας ως χώρα, κάτι που αναφέρθηκε πολλές φορές ε, σήμερα. Όμως θέλω να υπογραφήσω ότι το δικό μας φορολογικό σύστημα έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει εγκριθεί και από τον ΟΣΑ. Κάτι το οποίο δεν αναφέρθηκε εδώ από τους προλαλήσατες που αναφέρθηκαν στη χώρα μου. Επίσης, εμείς είμαστε κατά της φοροαποφύγης, όμως έχουμε κάποιες επιφυλάξεις σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος αυτού κοινή φορολογικής βάσης επιχειρήσεων. Και υπάρχει μια αιτιολογημένη γνώμη από το Κοινοβούλιο της Μάλτας επ' αυτού. Και εκεί αναφέρονται διάφορα μέτρα τα οποία πλήττουν την αρχή της επικουρικότητας. Όπως, για παράδειγμα, η κοινή φορολογική βάση επιχειρήσεων είναι εθελοντική στην περίπτωση επιχειρήσεων που δεν έχουν το χρόνο πάνω από 650 εκατομμύρια. Και έτσι θα υπάρχουν διαφορετικές προδιαγραφές. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα οι χώρες μέλη να πρέπει να αλλάξουν το φορολογικό του συντελεστή, με το οποίο δεν συμφωνούμε. Εμείς πιστεύουμε ότι η φορολόγηση είναι κυρίαρχο δικαίωμα της κάθε χώρας μέλος. Συνεπώς, πιστεύουμε ότι η επιλογή πρέπει να μείνει στις χώρες μέλη για να επιτεθούν οι στόχοι που βρίσκονται πίσω από την κοινή φορολογική βάση επιχειρήσεων. Χωρίς παρέμβαση στην αρχή της επικουρικότητας και αναλογικότητας. Έχουμε και επιφυλάξεις για την ίδια την διατύπωση, γιατί πιστεύουμε ότι θα οδηγήσει σε απώλεια εσόδων εφόσον γίνει φορολόγηση στην χώρα προορισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος την ε, Γαλλική Εθνοσυνέλευση και στη συνέχεια Δανία. Ευχαριστώ. Ναι, θα είμαι σύντομος, λέει ο κύριο Σεμπλέ. Όλοι γνωρίζουμε ότι γίνεται συζήτηση και ότι υπάρχουν αποκλήσεις μεταξύ των χωρών μελών για το πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα της φορολογικής συνεισφοράς των ψηφιακών επιχειρήσεων αν πρέπει να υπάρχει διαφορετική μεταχείριση ή αν πρέπει μέσω του άξις να χειριστούμε αυτό το ζήτημα, κάτι το οποίο θα μας βοηθούσε μέσω πρόθεσμα να καταλήξουμε. Όσον αφορά τη Γαλλία λοιπόν, εμείς υποστηρίζουμε μια διακριτή μεταχείριση και σύντομη. Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε πού έχει καταλήξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επ' αυτού. Να που γνωρίζουμε ότι ετοιμάζεται νομοθετική πρόταση που θα υποβληθεί τέλη Μαρτίου. Υπάρχουν ε, κάποιες θέσεις που έχετε καταλήξει στην διακριτή μεταχείριση ή μέσω του άξης. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Τέλφοντ, Δανία τώρα. Και μετά ο κύριος Πόρτεν, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζω να μπορέσουμε να ακούσουμε απάντηση στην ερώτησή σας. Το μεγαλύτερο τμήμα της νομοθεσίας που συζητούμε εδώ δεν είναι απαραίτητα κατανοητό για τους ε, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον τους περισσότερους εξ αυτών. Είναι πάρα πολύ σύνθετο και φυσικά δεν θα πρέπει να περιμένουμε να το κατανοήσουν, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Αλλά ένα εξ αυτών είναι και νομίζω ότι θα πρέπει να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη ε, των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι η μαύρη λίστα. Και κατά την άποψή μου δεν λειτουργεί η μαύρη λίστα. Ε, είναι μια ιδέα. Είναι ανεπαρκής και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν θα μπορέσει να αποκαταστήσει και την εμπιστοσύνη των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στα ε, θεσμικά όργανα που αποτελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε κάποια ένδειξη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διατεθειμένη να δημιουργήσει έναν αξιόπιστο τρόπο να παραμένουν τα χρήματα στις χώρες μας και να αντιπαλέψουμε αυτές τις πολυεθνικές επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή ε, μας εξαπατούν και δημιουργούν αυτές τις ανισότητες. Θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Πολ Τάγκ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μετά η κυρία Πέρετς από την Κροατία. Βλέπω κάποιους από τους αδέλφους που συνάντησα στη Γαλλία και στην Ιρλανδία, έχω τον κύριο Βόλκαν εδώ, από τότε που Αλένο Λαμασούρ, ο συνεισηγητής και εγώ, ε, ταξιδεύουμε ανά την Ευρώπη για να δούμε και τι έχουν να συμβάλλουν τα Εθνικά Κοινοβούλια για την κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση. Το Κοινοβούλιο θα εγκρίνει, ελπίζουμε αυτή την εβδομάδα στην Επιτροπή και το Μάρτιο στην Ολομέλεια την πρώτη ανάγνωση του κειμένου και ε, ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να ε, εξυγχρονίσουμε τα ε, επιχειρηματικά φορολογικά συστήματα. Είναι παροχημένα. Είναι από τότε που είχαμε υψικαμίνους στα εργοστάσια και επομένως αυτή τη στιγμή ε, πρέπει ε, να δούμε τι γίνεται με τις επιχειρήσεις, η οικονομική τους δομή, ε, αποφασίζουν ουσιαστικά πού θέλουν να κάνουν κέρδη και πού να φορολογούνται. Και η ενοποιημένη φορολογική βάση το αντιστρέφει. Οι επιχειρήσει θα αποφασίζουν πού θα πληρώνουν φόρου, πού θα έχουν το κύκλο εργασιών του ε, οι επιχειρήσει. Αυτό είναι το πρώτο και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να τροποποιηθεί η πρόταση για να συμπεριλάβει και τη φορολόγηση τη ψηφιακή οικονομία. Και νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτιμά μια διαρθρωτική λύση. Ε, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ανάγκη να φορολογηθούν οι ε, ε, γίγαντες αυτής της ψηφιακής οικονομίας. Από την άλλη όμως η έμεση φορολόγηση θα μπορούσε να υπάρχει βραχυπρόθεσμα, αλλά το διαρθρωτικό είναι να το περιλάβουμε στην άμεση φορολόγηση και να το εντάξουμε στο φορολογικό σύστημα. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξει ο ορισμός, ο ορισμός της μόνιμης εγκατάστασης, γιατί αυτό εκμεταλλεύονται οι Amazon και οι υπόλοιποι τώρα για να μην πληρώνουν φόρους. Επίσης, δεν γίνεται να μην περιμένουμε τον ΩΣΑ. Υπάρχει σαφή σύγκρουση συμφορών των μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο ΩΣΑ μπορεί να προχωρήσει μόνο αν η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλάβει τα ενία. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρησιμοποιούμε τα όσα κάνει ο ΩΣΑ, ε, χρησιμοποιούμε τα όσα κάνει το προσωπικό για να τα συμπεριλάβουμε στις ε, συμβουλές μας. Υπάρχει δουλειά, δεν υπάρχει πολιτική βούληση ακόμα στον ΩΣΑ. Ευχαριστώ η κυρία Πέριτς από την Κροατία και στη συνέχεια ο κύριος Φέλτεν από τη Σουηδία. Η Κροατία υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά αυτές τις δημοθετικές προτάσεις, ιδίως όσον αφορά τη φορολόγηση της ψηφιακής ε, οικονομίας. Η Κροατία είναι υπέρ της ε, σταθερής ε, φορολογικής ε, έδρας των επιχειρήσεων. Είμαστε υπέρ των νέων προτάσεων της Κομισιόν. Βεβαίως πρέπει όλα αυτά, όλες αυτές οι έννοιες να αποσαφινιστούν με σαφείς ορισμούς. Επίσης η Κροατία υποστηρίζει τη δυνατότητα να εξεταστεί το ενδεχόμενο να θεσπιστεί κοινό φορολογικό συντελεστή για τους διαδικτυακούς γίγαντες ώστε να γίνεται δυνατός ο έλεγχος των κερδών τους και να γίνεται δυνατή το να σχηματιστεί μια σαφής εικόνα για το τελικά, ποιο είναι τελικά το ύψος των κερδών που αποκομίζουν οι εταιρείε αυτές από την δραστηριότητά τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες που έχουν προταθεί θεωρούμε ότι μπορούν να συμβάλλουν στην μακροπρόθεσμη ε, επίλυση των προβλημάτων που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ ο κ. Φέλτεν από την Σουηδία και συνέχεια ο κ. από την Αυστρία. Ευχαριστώ πολύ. Με το έργο του ΟΣΑ για τα BEPS ε, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμβαδίσει με, αυτά τα έργα, με αυτό το έργο του ε, ΩΣΑ ώστε να το, επιληθούν τα προβλήματα της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής και είναι σημαντικό σε, ε, ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουμε σαφή εικόνα για το ποιοι είναι οι στόχοι προκειμένου να μπορέσουμε να τους επιτύχουμε από κοινού και συλλογικά. Θα πρέπει να έχουμε αντίληψη και επίγνωση του γεγονότος ότι αποτελούμε το, ε, ένα μέρος ε, της παγκόσμιας κοινότητας, του κόσμου ολόκληρου και γι' αυτό θα πρέπει με μια ενιαία φωνή να εμφανιστούμε στα διεθνή φόρα πρέπει να ε, εσωτερικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμφωνήσουμε επί των ορισμών που θα χρησιμοποιηθούν στις, ε, στις νομικές πράξεις που θα αποφασιστούν γιατί αυτά θα επηρεάσουν και, το γίγνεσθε στις άλλες χώρες. Το ερώτημά μου προς την Επιτροπή είναι έχετε σκοπό να δουλέψετε σκληρά προς αυτή την κατεύθυνση και τι μέτρα προτίθεστε να πάρετε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ρόσμαν από την Αυστρία και ο κύριος Κάρτη από το ΕΛΚ θα είναι ο τελευταίος μας ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι τα τελευταία χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη την καταπολέμηση φοροποφυγής και φοροδιαφυγής έγιναν πολλά, αλλά δυστυχώς πολλές φορές επεδείχθη επιφυλακτικότητα, ενώ πολλά ζητήματα παραμένουν ανοιχτά. Ε, είναι χαρακτηριστικό ότι το, τα, τα εθνικά αλλά και το διεθνές δίκαιο όσον αφορά τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας βρίσκονται ακόμα στη λίθινη εποχή. Θα ήθελα λοιπόν ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να μας πει αν έχει επεξεργαστεί η υπηρεσία του προτάσεις για αυτό το θέμα ε, τι πιστεύετε για παράδειγμα για τη δημιουργία ενός μηχανισμού για την παρακολούθηση και τη φορολόγηση των ψηφιακών εταιρεών ταυτόχρονα η διαφάνεια είναι ένα από τα σημαντικότερα ε, όπλα που έχουμε στη φαρέτρα μας για την καταπολέμηση φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής ωστόσο και εδώ επεδείχθη τεράστια επιφυλακτικότητα και υποχωρητικότητα αυτό αφορά και τα tax rulings και τις συστάσεις αναχώρησης αλλά και την τέταρτη οδηγία για την ε, καταπολέμηση της ε, νομιμοποίησης παράνομων εσόδων όπου δεν τελικά κατέστη δυνατό να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια στον τομέα των ιδρυμάτων και των ε, συλλόγων. Δημόσια πρέπει να είναι όλα τα στοιχεία διαφανή. Τίποτα λιγότερο. Και τέλος, μαύρη λίστα φορολογικών παραδείσων που καταρτίστηκε από το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών. Δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι δεν έχει καμία απόλυτη αξία μια τέτοια μαύρη λίστα αν σε αυτήν δεν μπορούν να συμπεριλαμβάνονται και ευρωπαϊκές χώρες. Κύπρος, Μάλτα, Ιρλανδία για παράδειγμα και ε, ιδίως οι Ηνωμένε Πολιτείε της Αμερικής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν, ο τελευταίος ε, ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ τους προσκεκλημένους μας. Είναι σαφές από τη συζήτηση μέχρι τώρα ότι υπάρχουν ε, διαφορές μεταξύ των Ευρωπαίων ε, εκπροσώπων και των εθνικών βουλευτών, των ευρωβουλευτών και των εθνικών βουλευτών για το πού ξεκινάει και πού τελειώνει η φορολογική κυριαρχία. Το ξέρουμε αυτό από τις διάφορες προτάσεις που έγιναν για την κοινή φορολογική βάση επιχειρήσεων κλπ. Όμως, ως εκλεγμένοι, αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει είναι η διαφάνεια. Ο κύριος Λάγκε στην έκθεσή του λέει ότι η Ερευνητική Επιτροπή για τα Panama Papers που δημιουργήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρέθηκε αντιμέτωπη με πάρα πολλά εμπόδια και από την Επιτροπή και από το Συμβούλιο προκειμένου να μπορέσουν οι ευρωβουλευτές να έχουν πρόσβαση στα διάφορα έγγραφα. Εδώ λοιπόν είναι θέμα κώδικα θετολογίας του Συμβουλίου όταν πρόκειται για τα φορολογικά. Άρα λοιπόν πρέπει εδώ να ακολουθήσουμε κοινή γραμμή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια, να συνεργαστούμε στο μέλλον προκειμένου να αναγκάσουμε αυτούς που δεν θέλουν να λογοδοτήσουν, να λογοδοτήσουν απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες. Οι εθνικοί βουλευτές δηλαδή εδώ έχουν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο γιατί μπορούν να επηρεάσουν τις κυβερνήσεις τους. Και εμείς από την πλευρά μας έχουμε πολύ σημαντικό ρόλο γιατί μπορούμε να επηρεάσουμε την Επιτροπή και το Συμβούλιο για να υπάρξει διαφάνεια επιτέλους όσον αφορά τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Συλλογικά λοιπόν πρέπει να φροντίσουμε για να δημιουργηθεί επιτέλους ένα σύστημα φορολογικής δικαιοσύνης. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Έχει τελειώσει περίπου ο χρόνος μας, αλλά θα δώσουμε το λόγο στους κύριους ομιλητές μας εδώ για να απαντήσουν όσον αφορά τις προτάσεις που κάνανε και τις ερωτήσεις που ακολούθησαν. Παρακαλώ, ο κύριος Μουτρελιέ. Ευχαριστώ πολύ. Σε ένα λεπτό, ναι, θα προσπαθήσω να απαντήσω, είναι βέβαια δύσκολο. Για τα τέλη Μαρτίου ετοιμάζουμε ένα πακέτο προτάσεων για να φορολογηθούν καλύτερα οι ψηφιακές επιχειρήσεις. Δηλαδή θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τα έσοδά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί όπου τα προσωπικά δεδομένα οδηγούν στην δημιουργία εσόδων. Και αυτό ε, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΣΑ. Κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε μία πρόταση που να επικεντρώνεται βραχυπρόθεσμα, ώστε περιμένοντας τις διαπραγματεύσεις να καταλήξουμε αργότερα ε, σε κάτι μακροπρόθεσμα. Τώρα για τον ε, δικό μας κατάλογο. Αυτό που έχει σημασία είναι τα αντίμετρα. Πάνω σε αυτά οι χώρες μέλη δεν έχουν προχωρήσει. Εμείς θέλουμε να μην δίνονται κονδύλια στις επικράτες εκείνες όπου δεν συμμορφώνονται. Επίσης θέλουμε να είναι δημόσια τα δεδομένα και αυτό θέλουμε οι νομοθέτες να το εγκρίνουν και θα έπρεπε ο κατάλογος των επικρατείων αυτών που δεν συνεργάζονται να είναι δημόσιος, γιατί μόνο τότε θα υπάρξουν αλλαγές. Όσον αφορά τώρα την ε, κυριαρχία και το άξις, εγώ ναι, να συζητήσω όσο ενδιαφέρονται το άξις, όπως έλεγε και ο κύριος Τάνκ, είναι για να ενισχύσει τη φορολογική κυριαρχία, προκειμένου δηλαδή οι για την, τον τόπο φορολόγησης να είναι κάτι που θα αναλάβουν οι δικήσεις. Και αυτό θέλουμε να το κάνουμε μαζί μέσα στην ενιαία αγορά. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Ε, πρέπει να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Οπωσδήποτε. Ωραία, 30 δευτερόλεπτα κύριε Λάγκεν. Για μια πολύ σύντομη παρατήρηση μόνο. Δύσκολο. Διαφάνεια είναι το σημαντικότερο. Όχι μόνο διαφάνεια μεταξύ των φορολογικών αρχών, αλλά και ως προς την ε, δημοσιοποίηση των ε, εμπορικών ε, και εμπορευματικών μεταφορών ή στις, στις εταιρείες ταχυδρομικές θερίδες. Δεύτερον, παραδείγματα που δεν συζητήσαμε είναι, που δεν συζητήσαμε είναι χρυσές θεωρήσεις, μεταφορές με πλοίο, εκεί υπάρχουν χώρες οι οποίες πρέπει να λάβουν πολύ συγκεκριμένα μέτρα κάτι που θα συζητήσουμε και θα εξετάσουμε στο πλαίσιο της τρίτης επιτροπής τάξε 3 που θα συστήσουμε και προσβλέπω και ελπίζω και στη δική σας συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα πλέπει ε, πραγματικά αν έχετε μία πολύ σύντομη, σύντομη παρατήρηση, διότι έχουμε τους καλεσμένους μας που πρέπει να μιλήσουν στο επόμενο πάνελ και δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε άλλο. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη σε όλους τους ομιλητές μας. Ε, είναι καλό σημάδι το γεγονός ότι υπάρχει ε, τόσο ενδιαφέρον και τη ζωτική σημασία στο θέμα για όλους μας. Πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί και προσβλέπουμε και στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, παρακαλώ, διαβάστε και την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση επιχειρήσεων. Τώρα περνάμε στο δεύτερο τμήμα, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό, η Τραπεζική Ένωση η διαχείριση της ε, ισορροπίας μεταξύ καταμερισμού κινδύνου και μείωσης του κινδύνου. Εύκολο θέμα. Και έχουμε εδώ και αξιότιμους προσκεκλημένους, όπως και στο προηγούμενο πάνελ. Ο πρώτος ομιλητής είναι καθοδόν ακόμα. Εν τω μεταξύ λοιπόν εγώ να σας πω ότι ε, ασχολούμαστε με το πακέτο τη δέσμη μέτρων για τα τραπεζικά θέματα, τη μείωση του κινδύνου, το CRR, το CRD και το BRRD και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τι εργασίε σε εγκαίρω ώστε να ξεκινήσει ο τριμερή διάλογο πριν από το καλοκαίρι και να ολοκληρώσουμε με το νομοθετικό θέμα αυτό πριν από το τέλο του έτου. Επιπλέον στοιχείο μείωση κινδύνου λοιπόν, ελπίζουμε να ολοκληρωθεί και αυτό. Περιμένουμε και τη δέσμη μέτρων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζουμε να τη διαβάσει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και φυσικά θα ακούσουμε και τον εισηγητή για το θέμα ε, έντις και ελπίζουμε να έχουμε και την παράλληλη διάσταση διότι όπως σας είπα το θέμα της, ε, του περιορισμού του κινδύνου θα αλλάξει, θα αλλάξει και το θέμα του καταμερισμού του κινδύνου, θα δούμε όμως, αυτό θα συζητήσουμε τώρα. Ο Ολιβιέ Κερσον, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης ΦΙΣΜΑ είναι εδώ. Συνάδελφοι, λίγο ησυχία παρακαλώ. Και αυτός και είναι ο πρώτος ομιλητής μας. Ολιβιέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Ρομπέρτο. Κυρίες και κύριοι, από το 2010 και μετά, η ιστορία της ε, χρηματοπιστωτικής επιπτείας και της χρηματοπιστωτικής ρύθμισης είναι γνωστή. Ε, πάνω από 50 νομοθετικά κείμενα παρουσιάστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ψηφίστηκαν και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά έχουμε υπόψη μόνο τις τράπεζες, στον τραπεζικό τομέα, αυξήσαμε ε, την αφαιρεγγιότητες ε, για τις τράπεζες, ε, δημιουργήσαμε επιπλέον δικλείδες ασφαλείας, υπάρχει μόχλευση, ποσοστά ρευστότητας και τροποποίησαμε και τη διακυβέρνηση αυτών των οργανισμών και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Αναφέρω απλώς κάποια από τα πολλά μέτρα που εγκρίθηκαν από αυτό το κοινοβούλιο στα πλαίσια του δέσμης μέτρων για τα θέματα αυτά. Επίσης υπήρχε το θέμα της εξυγίασης των τραπεζών απαιτήσει 8% ε, MRL πριν να υπάρχει πρόσβαση στα κονδύλια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχουμε ξεκινήσει την Τραπεζική Ένωση που εδράζεται σε τέσσερις πυλάνες. Ε, χρειαζόμαστε ένα κατάλληλο μηχανισμό. Από τον Νοέμβριο του 2014 ε, περάσαμε στο μηχανισμό εξυγίανσης, ο οποίος ε, ξεκίνησε να εφαρμόζεται ένα χρόνο αργότερα, ένα πρόγραμμα εγγυήσεων, το οποίο είναι προς εξέταση από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και ένα ε, κοινό backstop. Τα δύο πρώτα στοιχεία είναι ήδη σε εφαρμογή. Το backstop έχει συμφωνηθεί από τους Υπουργούς από το 2013 και θα τεθεί σε εφαρμογή το αργότερο στο τέλος της μεταβατικής περίοδου των 8 ετών. Όσον αφορά τον καταμερισμό κινδύνου, αυτή τη στιγμή έχουμε το θέμα του Ταμείου ε, Εξυγίανσης, ε, το οποίο θα προχωρήσει ε, και θα ολοκληρωθεί σε αυτό το εκταετές μεταβατικό πλαίσιο. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μεγάλη βελτίωση στις κεφαλαϊκές και ε, θέσεις ρευστότητας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής, ε, των Ευρωπαϊκών Τραπεζών. Θα προχωρήσουμε το τραπεζικό τομέα και θα θέσουμε σε ισχύ ένα μηχανισμό σημαντικής ενίσχυσης ε, της φερεγγιότητας των τραπεζιών. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ολοκληρώσαμε με τη μείωση του κινδύνου, σαφώς όχι. Το Συμβούλιο του Ιουνίου του 2016 κατάρτισε έναν οδικό χάρτη, ο οποίο εξακολουθεί να ισχύει πλήρω ακόμα και σήμερα, τουλάχιστον αυτό πιστεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και πιστεύει ότι ο καταμερισμό του κινδύνου θα πηγαίνει χέρι-χέρι με την μείωση του κινδύνου και αυτό ακριβώ κάναμε μέχρι τώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε το θέμα ε, το 2016 με διαδοχικές ε, επιτυχής προεδρίας και έχουμε ελπίδες ότι θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τριμερή διάλογο ε, την Άνοιξη με στόχο να ολοκληρώσουμε τη διαπραγμάτευση ή δυνατόν μέχρι τον Ιούνιο αλλά τουλάχιστον πριν από το τέλος του έτους. Έχουμε κρυζώσει τον κίνδυνο στο τραπεζικό σύστημα. Σε καμία περίπτωση βεβαίω, αλλά δεν θα πρέπει να είναι αυτό ο στόχο μα. Ε, τα τραπεζικά θέματα προϋποθέτουν και κινδύνους, γιατί αλλιώς είναι κάτι άλλο, δεν είναι τραπεζικά ζητήματα. Αυτό το οποίο κάνουμε και συνεχίζουμε να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε τις δυνατότητες των ε, τραπεζών να είναι καλύτερες εξοπλισμένες για να έχουν ένα καλύτερο σύστημα διαχείρισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επ' αυτή τη βάση, λοιπόν, είναι τη άποψη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η μείωση του κινδύνου και καλύτερα μέσα διαχείριση κινδύνου θα μα επιτρέψει να έχουμε κατάλληλο επιμερισμό και να έχουμε ε, μηχανισμούς όπως για παράδειγμα η περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας από τον κίνδυνα και αυτό φυσικά σημαίνει ότι θα βγουν κερδισμένοι όλοι. Να προσθέσω επίσης ότι αυτή τη στιγμή δεν ε, συμμορφόμαστε μόνο με τον οδικό χάρτη του 2016, αλλά έχουμε πάει και παραπέρα ε, από τα όσα ζητούνται. Όσον αφορά τα μέτρα για τη μείωση του κινδύνου που προβλέπονταν σε αυτό το χάρτη, ε, όπως μόλις ανέφερε ο πρόεδρος Γκουαλτιέρη, πολύ σύντομα θα έχουμε ένα ε, πακέτο για τα δάνεια που δεν εξυπηρετούνται, το οποίο δεν προβλεπόταν στον οδικό χάρτη, ε, το οποίο κατά την άποψή μας θα είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό για τη μείωση του κινδύνου. Πιστεύουμε ότι χρειάζεται δια, ε, επίουσα πρόοδος στο άλλο τμήμα του οδικού χάρτη, κυρίως ε, όσον αφορά τον επιμερισμό κινδύνου. Τον Οκτώβριο η ανακοίνωση για την Τραπεζική Ένωση ε, υπέδειξε κάποια λύση για ένα πιθανό συμβιβασμό και φυσικά ενθαρρύνω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προχωρήσει και να εγκρίνει όσο το δυνατόν ε, πιο σύντομα την έκθεση για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε και συγκεκριμένε διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο. Θα ήθελα να αναφέρω ότι η πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φαίνεται να ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις ιδέες ε, του ε, εισηγητή, τον οποίο θα ήθελα να συγχαρώ για την εξαιρετική δουλειά που έκανε σήμερα και φυσικά ε, το γενικότερο σκεπτικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, το έντις στο στάδιο 1 θα πρέπει να οδηγήσει σε βοήθεια ρευστότητα, δεν θα περιλαμβάνει όμως πλέον επιμερισμό κινδύνου. Κάτι το οποίο θεωρούμε ότι είναι και ένα από τα ε, δελεαστικά του στοιχεία και πρέπει να ληφθεί υπόψη και υπ' αυτή την άνοια έχουμε κάνει περισσότερα από όσα ζητούσε ο δικός χάρτης διότι αν συνεχίσουμε με αυτές τις ιδέες θα έχουμε ε, τουλάχιστον ελαφρά μικρότερο επιμερισμό κινδύνου, τουλάχιστον για την αρχή, και σημαντική μείωση του κινδύνου. Για να ολοκληρώσω λοιπόν, πρέπει να πιέσουμε, πιστεύω, για να έχουμε και το backstop, το δημόσιο backstop. Αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν, όλοι συμφωνούν ότι θα πρέπει να υπάρχει το backstop. Ε, όπως σας είπα συμφωνούν ε, οι υπουργοί, συμφώνησαν από το 2013 και όσο πιο σύντομα τεθεί σε εφαρμογή, τόσο πιο γρήγορα θα ε, σταθεροποιηθεί η Τραπεζική Ένωση και θα συμβάλλει αυτό και στη σταθεροποίηση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λοιπόν, ότι είναι σαφές ε, και είναι ζωτική σημασία ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση εντός της εντολής αυτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ε, πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας να το ολοκληρώσουμε αυτό τώρα ε, μετά από τον οδικό χάρτη του Προέδρου Τούσκ. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπράκμαν από την Bundestag. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, για την αφαιρεγιότητα των τραπεζών θέλουμε να ενισχύσουμε τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα των τραπεζών και να προστατευτούμε από την, ε, ε, από την απώλεια εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα από αυτή την άποψη ε, είναι σημαντικότερο να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός προστασίας των καταθέσεων. Αλλά όπως και σε όλους τους μηχανισμούς προστασίας πρέπει να εξασφαλιστεί ότι ε, αυτή η ασφάλιση δεν θα καλύπτει ε, κινδύνους και ρίσκα που υπάρχουν ήδη Όπω οι κίνδυνοι που έχουν αναλάβει ήδη οι τράπεζες και επίσης ότι δεν θα μπορούν να καλύψουν ε, δυσανάλογα πολύ ε, ε, τους κινδύνους που θα αντιμετωπίσουν οι τράπεζε στο μέλλον. 60 ε, δισεκατομμύρια είναι τα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι υπερβολικά πολύ. Γι' αυτό και όρος για τη δημιουργία ενός μηχανισμού προστασίας είναι να μειωθούν σημαντικά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αυτό είναι απαραίτητος όρος για τη δημιουργία του μηχανισμού προστασίας και εγγύηση των καταθέσεων. Δεν θα μπορέσει να γίνει δεύτερο ή τρίτο βήμα αν ε, δεν ε, απομειωθούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο παρόν, αλλά και αν δεν αποκλειστεί μια παρόμοια εξέλιξη και στο μέλλον όσον αφορά τη συσσόρευση τέτοιων μη εξυπηρετούμενων δανείων. Χρειάζεται λοιπόν μια αναδιάρθρωση των τραπεζών, αλλά θα πρέπει να μειωθεί ε, το επίπεδο του κινδύνου και να καταρτιστούν σοβαροί, αυστηροί κανόνες ακριβώς για να αποφεύγονται τέτοια φαινόμενα στο μέλλον. Το, πόσο, ε, το πόση δουλειά ε, θα πρέπει να γίνει αποτυπώνεται και στη σχετική έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν θέλω να θέσω το ερώτημα αν η ΕΚΤ υπερεύει τις αρμοδιότητες του, τις αλλά θα περιμένω τις κατευθύνσεις γραμμές που θα εκδώσει τον Μάρτιο. Όμως ε, προειδοποιώ ε, όσον αφορά τον κίνδυνο να αποδυναμηθούν οι κανόνες που θα θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αντίθετα λοιπόν από την αποδυνάμωση χρειαζόμαστε ενιαίους αυστηρούς κινδύνους τόσο όσον αφορά τη χορήγηση δανείων, αλλά όσο και όσον αφορά την ε, διαχείριση των κινδύνων που ε, προκαλούνται αναγκαστικά και αντικειμενικά από τη χορήγηση δανείων. Τέτοιοι κανόνες υπάρχουν σε πολλές χώρες και στη Γερμανία. Ε, βασικό στοιχείο είναι η κατά προτεραιότητα διαχείριση και αντιμετώπιση του δημόσιου χρέους. Τέτοιοι κανόνες πρέπει να καταργηθούν. Ε, τα δάνεια σε δημόσιους φορείς δεν είναι ε, δάνεια χωρίς κίνδυνο και χωρίς ρίσκο. Η ίδια η κρίση που ε, ξέσπασε πριν από 10 χρόνια απέδειξε ακριβώς αυτό. Τα χρεόγραφα και τα ομόλογα που εκδίδονται από, την, ε, από τα κράτη αλλά και τα ευρωομόλογα όπως έχουν προταθεί δεν αποτελούν ε, λόγο για την αποδυνάμωση των, ε, κανόνων που έχουν ήδη θεσπιστεί. Τα δάνεια που κατευθύνονται σε δημόσιες φορείς δεν θα πρέπει να διέπονται από διαφορετικούς κανόνες σε σχέση με εκείνους που ισχύουν για τους ιδιώτες. Ξέρω ποιες είναι οι προτάσεις και ποιες είναι τα, ποια θα ήταν τα αποτελέσματα μιας τέτοια στάσης όπως αυτή που περιγράφω και ξέρω πόσες αντιδράσεις ενδέχεται να προκληθούν. Όμως χρειαζόμαστε μια ενιαία ανθεκτική τραπεζική ένωση και κατά την οικοδόμησή της χρειάζεται να αποφύγουμε προβλήματα που έχουν εμφανιστεί στο παρελθόν και που τα έχουμε διαπιστώσει όλοι από κοινού. Δεν είναι δυνατόν να διατρέξουμε τον κίνδυνο να καταρρεύσει ολόκληρο το οικοδόμημα αυτού που πάμε να χτίσουμε, ακριβώς γιατί τα θεμέλια που θα έχουμε θέσει θα είναι πολύ αδύναμα. Ευχαριστούμε κύριο Βανσάν Εμπλέ, λοιπόν, από την Επιτροπή Οικονομικών της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ πρώτα απ' όλα τους προλαλήσαντες. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ σε αυτήν την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ εθνικών βουλευτών και ευρωβουλευτών παρόλο που εμείς υποδεχτήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα μια αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι επαφές αυτές είναι πολύτιμες γιατί εμπλουτίζουν τον προβληματισμό μας. Με την Τραπεζική Ένωση λοιπόν και με την ανάληψη των κινδύνων κάνουμε μια δοκιμή της ικανότητας των χωρών από κοινού να αναλάβουν τους κινδύνους. Βέβαια πολλά ερωτήματα τίθενται ε, και τα έχει ήδη εκφράσει η Γαλλική Γερουσία από το 2012. Μιλήσαμε για την ε, ενιαία εποπτεία και η Γερουσία μας ενέκρινε τη σχετική ευρωπαϊκή πρόταση. Στη συνέχεια έκανε διάφορες προτάσεις για βελτίωση αυτού του πρώτου πυλώνα. Η Επιτροπή Οικονομικών μας επέμεινε κυρίως για τρία πράγματα. Πρώτον, να συμπεριληφθεί η διασφάλιση μέσα στην εποπτεία. Δεύτερον, εναρμόνιση των εθνικών διαδικασιών εξυγίανσης που για μας έπρεπε να είναι προϋπόθεση για να αρχίσει να ισχύει ο ενιαίος μηχανισμός. Και τρίτον, απαιτήσαμε την συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων στην εποπτεία. Και η διάσκεψη που προβλέπεται από το άρθρο 13, βάσει της οποίας βρισκόμαστε και εδώ σήμερα, θα έπρεπε ακριβώς αυτό το ρόλο να επιτελεί. Όσον αφορά τώρα το δεύτερο πυλώνα της Τραπεζικής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα το ενίο ταμείο εξυγένσης ήταν κάτι που συζητήθηκε στη Γερουσία μας και το 2015 υιοθετήσαμε τροπολογία για τον ενίο αυτό μηχανισμό και τον εξαρτήσαμε από την επικύρηση του διακυβερνητικού ορισμού ο, η γερουσία μας δηλαδή ήθελε έτσι να δείξει το ενδιαφέρον του για την ανακράτος αντιμετώπιση μέχρι να υπάρξει αυτός ο επιμερισμός. Αυτό αντικατοπτρίζει την ανησυχία μας όσον αφορά την εισφορά της Γαλλίας στο ταμείο αυτό το κοινό επίλυσης. Η συνεισφορά αυτή θα σήμαινε λιγότερα χρήματα για την γαλλική οικονομία. Και ο Υπουργός Οικονομικών στήριξε τον μηχανισμό, κρούντας όμως τον κόδωνα του κινδύνου. Εδώ και δύο χρόνια λοιπόν γίνονται ξανά και ξανά συζητήσεις για το σύστημα εγγύσεων καταθέσεων. Και τον Μάρτιο του 2016 ακούσαμε την κυρία Κενίκη, πρόεδρο του ενιαίου ταμείου. Και στην ανταλλαγή αυτή απόψεων εμείς υπογραμμίσαμε ότι η επίλυση αυτή των τραπεζών αποτελεί μια πρόοδο γιατί είναι οι μέτοχοι εκείνοι οι οποίοι πρώτα πρέπει να επομίζονται τις απώλειες. Και γι' αυτό και η Γερουσία τότε είπε ότι τα μαθήματα από την οικονομική κρίση του 2008 ήταν μαθήματα που είχαμε μάθει. Τώρα, σε περίπτωση ε, απώλειας πρέπει να υπάρξει εξυγίανση και όχι εκαθάριση και να υπάρχει ένα Ταμείο Εθνικών που είναι υποχρεωτικό από τις 30 Μαΐου του 2014. Και έτσι έρχομαι στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύσεων Καταθέσεων, που είναι ο τρίτο πυλώνας τη Τραπεζική Ένωση. Η εγγύηση καταθέσεων διχάζει τις χώρε μέλη. Η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μάλιστα έχει εξελιχθεί με το χρόνο. Το 2016, για παράδειγμα, η Γερουσία είχε χαιρετήσει την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κάποιε επιφυλάξει. Η αρχική πρόταση έλεγε ότι πρέπει να γίνει παραπάνω προσπάθεια με 7 δισεκατομμύρια από πλευρά των γαλλικών τραπεζών για να καλυφθεί ε, περισσότερο η κατάσταση από τη μέχρι τότε. Και η Γερουσία σκέφτηκε ότι αν αυτή η εγγύηση καταθέσεων κερδίζει σε αξιοπιστία στα μάτια των πολιτών, από την άλλη μεριά ο τρόπος χρηματοδότησης πρέπει να εξαρτάται από τον κίνδυνο. Στη συνέχεια η Γερουσία συμφώνησε με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ότι η Τραπεζική Ένωση δεν μπορεί να λειτουργήσει παρά μόνο εφόσον ε, υπάρχει μείωση του κινδύνου. Και για να έρθω σε αυτά που είπα και οι συνάδελφοι, η Τραπεζική Ένωση ε, απαιτεί να τακτοποιηθεί το θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Είναι και αυτό θέμα προτεραιότητας. Η μείωση του κινδύνου πρέπει να πάει παράλληλα με την εγγύηση καταθέσεων. Είναι κάτι που επιθυμούμε βέβαια να γίνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Πάολο Γκαριέρη από την Ιταλική Γερουσία τώρα. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω καταρχάς είναι σημαντικό να πούμε ότι η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης είναι ουσιώδες βήμα προκειμένου να μειώσουμε τον ε, ε, οικονομικό κατακαιρματισμό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή στην Ευρωζώνη. Επίσης ε, πρέπει να δούμε και ε, αυτούς τους καρχαρίες που έχουμε στον ευρωπαϊκό χώρο. Χρειάζεται λοιπόν μια ουσιαστική αναγνώριση που πρέπει να κάνουμε ευθύ εξ αρχή. Η ολοκλήρωση της τραπεζικής άνωση θα δώσει και μεγαλύτερο ρόλο στο ιδιωτικό κεφάλαιο για να μπορέσει να, να μετριάσει ε, τα χρηματοπιστωτικά σόκο. Και ακούγοντας και την προηγούμενη παρέμβαση, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι η μόνη βιώσιμη λύση είναι να βρούμε κάποια ικανοποιητικό συμβιβασμό μεταξύ αυτών των δύο αναγκών. Αφενός ε, την ε, μείωση του κινδύνου στα τραπεζικά ισοζύγια και ταυτόχρονα να έχουμε κατάλληλο επιμερισμό κινδύνων. Ε, είναι σαφές ότι ο κίνδυνος ε, προκύπτει από το μεγάλο αριθμό μη εξυπηρετούμενων δανείων και την έκθεση των τραπεζών ε, στην εθνική τους κυριαρχία. Όσον αφορά τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καταρχάς θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι γίνονται ήδη σημαντικές προσπάθειες. Στην περίπτωση, για παράδειγμα, της Ιταλίας, ε, η προληπτική κεφαλαιοποίηση της τράπεζας Μαντεπάσκη και δύο μικρότερων ε, τραπεζών και δύο μεσαίου μεγέθους τραπεζών θα οδηγήσουν σε μείωση κατά ένα τέταρτο ε, την τρέχουσα χρονιά. Ε, περαιτέρω πρόοδο στον τομέα αυτό κατά πάσα πιθανότητα θα, μειώσει, θα προκύψει και από μια πολιτική που ξεκινά από τον νέο μηχανισμό εποπτείας, ε, τα οποία βέβαια ακόμα πρέπει να τα καθορίσουμε καλύτερα. Αλλά από την άλλη η οικονομική ανάπτυξη κατά πάσα πιθανότητα θα διευκολύνει και τη μείωση των ε, μη εξυπηρετούμενων δανέων γιατί πολλές χρεοκοπημένες εταιρείε θα μπορέσουν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους. Η μείωση ε, επίσης ε, στα τραπεζικά χαρτοφυλάκια απαιτεί περαιτέρω δράση και σημαίνει ότι θα πρέπει να μειώσουμε την ε, προληπτική πολιτική μεγάλης έκθεσης, αλλά θα εξασφαλίσει και μια σταδιακή είσοδο με κατάλληλη στάθμιση των διαφόρων ε, κινδύνων για να μειώσουμε τις αρνητικές συνέπειες. Ορισμένες φορές η διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων θα ευνοείται και θα απαιτεί ε, και τη δημιουργία ενός μηχανισμού ευρωπαϊκού στοιχείων ενεργητικού που θα βοηθήσει να κάνουμε αυτή τη διαφοροποίηση. I think Πιστεύω ότι οποιαδήποτε άμεση ε, αξιολόγηση του κινδύνου της εθνικής κυριαρχίας γιατί μπορεί να επηρεάσει την αγορά της χώρας αυτής και τελικά θα δημιουργήσει περαιτέρω αστάθεια. Στο δεύτερο μέτωπο που είναι ο ευρύτερος επιμερισμός των κινδύνων νομίζω ότι θα μπορούσαμε να επιχειρηματολογήσουμε υπέρ ενός ευρωπαϊκού συστήματος ε, εγγύησεων ε, καταθέσεων και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει τέτοια πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να την υποστηρίξει, διότι θα είναι και ένας ικανοποιητικός συμβιβασμός για να έχουμε καλύτερο επιμερισμό κινδύνων όταν θα υπάρχει δημοσιονομικό backstop ε, μεταξύ των κονδυλίων. Στο πρώτο στάδιο, θα υπάρχει μία γραμμή πίστοσης ρευστού στα εθνικά προγράμματα τα οποία έχουν εξαντλήσει τους πόρους τους. Η συνεχής μετάβαση, ακόμα και σε μερική αμεβεοποίηση, μπορεί ε, να υπόκειται σε αποτελεσματική πρόοδο στη μείωση του κινδύνου και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αναγνωρίσουμε. Επίσης, δεν μπορούμε να σταματήσουμε σε αυτή τη διαδικασία του, της μόνο. Θα πρέπει ε, να γίνει πολλή δουλειά ώστε να μπορέσουμε να διασκεδάσουμε και τις ανησυχίε και για τον ε, ε, ε, βασικό κίνδυνο που υπάρχει, αλλά και για τον ηθικό κίνδυνο, το moral hazard. Θα πρέπει να υπάρχουν σημαντικές πολιτικές για να μειώσουμε το υπερβολικό ε, δημόσιο χρέος ε, με κατάλληλη αναλογία και πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε ένα καλύτερο σύστημα περιορισμών στον προπολογισμό στην εθνική δημοσιονομική πολιτική. Και έτσι θα ενισχύσουμε και θα έχουμε πιο αποτελεσματικούς κανόνες για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Πρέπει να αποφύγουμε όμως οποιαδήποτε αυτοματή ή μη αυτόματη διαδικασία αναδιάρθρωσης του χρέους ή τέτοια πρόταση του εθνικού χρέους, διότι πιστεύω ότι αυτό ε, υποβοηθά ε, τον κίνδυνο ε, δημοσιονομικής αστάθειας και θα την τροφοδοτήσει περισσότερο. Να συνοψίσω λοιπόν και να πω εν τέλει ότι πιστεύω ότι η τεχνική συνιστός μιας βιώσιμης συμβαστικής λύσης για να έχουμε την Τραπεζική Ένωση υπάρχει αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται και η κατάλληλη πολιτική βούληση. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμό για να ολοκληρώσουμε την Τραπεζική Ένωση και να είναι απεδεικτό αυτό από όλε τι πλευρέ ε, προ όφελο όχι μόνο τη τραπεζική σταθερότητα τη Ευρωζώνη αλλά και των πολιτών μα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Συμπρόεδρος έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γκουαλτιέρη. Νομίζω ότι μόλις ένα λεπτό μου μένει. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι ο επιμερισμός και η μείωση του κινδύνου είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Είναι βεβαίως λογικό το ότι επικεντρωθήκαμε περισσότερο στον ε, επιμερισμό του κινδύνου, όμως και τα δύο θέματα είναι απόλυτη ζωτική σημασία για τη σταθερότητα του τραπεζικού μας συστήματος αλλά και για την κοινωνικο-οικονομική εξέλιξη και ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Βουλγαρία και η Βουλγαρική Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έχουν ως στόχο να καταλήξουμε σε έναν αποδεκτό συμβιβασμό στα δύο αυτά θέματα. Θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας επί της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ώστε να εφαρμοστεί το έντις ε, κάτι που θα αποτελέσει με τη σειρά του και την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος. Και ξεκινούμε τώρα τις παρεμβάσεις των συναδέλφων. Η κυρία Λουκουκέρκ έχει το λόγο. Δύο λεπτά από την Πορτογαλία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να τοποθετηθώ. Καταλαβαίνω ότι έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο. Εγώ ήμουν στο Eurogroup και στο ECOFIN 2011-2015 και πράγματι υπήρχε μια περίοδος όπου σημειώσαμε πάρα πολύ γρήγορη πρόοδο όσον αφορά την θέσπιση μέτρων για την αντιμετώπιση των, της ε, κρίσης. Και πολλές από τις ιδέες που ακούστηκαν σήμερα τις είχαμε συζητήσει και εκείνη την περίοδο, 2011-2015. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι ο πρώτος στόχος είναι η μείωση του κινδύνου και ε, ε ταυτόχρονα αυτό να συνοδευτεί από επιμερισμό του κινδύνου. Όμως ανησυχώ ε, όσον αφορά τον μηχανισμό προστασίας και εγγύησης των καταθέσεων. Ελπίζω ότι δεν θα χρειαστεί άλλη μια κρίση ε, ώστε να καταλήξουμε και σε αυτό το στάδιο. Χρειαζόμαστε ε, τραπεζική ένωση, πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα και αυτό θα βοηθήσει στην ενίσχυση της σταθερότητας και της αξιοπιστίας του χρηματοπιστωτικού τομέα. Για πάρα πολλά χρόνια βλέπουμε να υπάρχουν πάρα πολύ χαμηλά επιτόκια αυτό με ταυτόχρονη ε, ε, ύπαρξη πολύ κανόνων και περιορισμών ε, έχει πλήξει σοβαρά την κερδοφορία των τραπεζών. Αυτό έχει οδηγήσει με τη σειρά του σε διακοπή της δανειακής ροής, της χορήγησης δανείων προς επιχειρήσεις. Ίσως λοιπόν έχει έρθει πλέον η ώρα να εξετάσουμε ενδεχομένως έναν νέο τραπεζικό κανονισμό, στον οποίο όμως θα έχουμε εκ των προτέρων ε, αξιολογήσει και αναλύσει τον κίνδυνο και τις επιπτώσεις, προκειμένου να, μην, ε, να, να αναιρεθεί και να καταργηθεί αυτό το πρόβλημα της ε, χρηματοδότησης των επιχειρήσεων από τις, από, τράπεζες. Ο κύριος Χαράγκα από τη Φιλανδία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως φαίνεται και στο Συμβούλιο και εδώ υπάρχει μεγάλη διαφωνία ε, ως προς το κατά πόσο έχουμε προσεγγίσει το στόχο της Τραπεζικής Ένωσης. Μπορούμε να συζητούμε τον, τον ορισμό ε, του επιμερισμού, της μείωσης του κινδύνου και όλων αυτών των όρων για πολλά χρόνια. Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να βάλουμε διαρκώς αυτή τη μεταρρύθμιση και ιδίως την Ένωση Κεφαλαιογορών που συνδέεται με την Τραπεζική Ένωση. Μήπως λοιπόν θα έπρεπε να, να υιοθετήσουμε μια διαφορετική προσέγγιση. Γιατί να μην υπάρχει μια συμμαχία προθύμων ή και των ικανών. Εκείνων δηλαδή που ε, συμφωνούν ότι η μείωση κινδύνου ε, είναι ε, απαραίτητη και επαρκής μπορούν να προχωρήσουν και στον επιμερισμό και με βάση τα θετικά αποτελέσματα που ενδεχομένως θα έρθουν να ε, ακολουθήσουν και ε, άλλες ε, χώρες αργότερα γιατί ε, όταν θα αρχίσει η συνεργασία και ο επιμερισμός κινδύνου όσον αφορά την, τους τραπεζικούς ισολογισμούς ε, και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και αφού θα έρθουν θετικά αποτελέσματα, αυτό θα αποτελέσει το καλύτερο κίνητρο και για όσους αυτή τη στιγμή προβάλλουν επιφυλάξεις και, και αντίσταση. Ξέρω ότι δεν θα είναι η καλύτερη ή πιο εύκολη λύση, αλλά νομίζω ότι θα είναι η πιο αποτελεσματική. Ευχαριστώ, κύριος Λάγκε. Η, κυρία Λάγκε. Ευχαριστώ, δεν το περίμενα. Ευχαριστώ πάντως, Πρόεδρε. Οι παρεμβάσει που ακούσαμε και από τους κύριους ομιλητές, αλλά και τα σχόλια από την αίθουσα, δείχνουν πόσο ευαίσθητο είναι αυτό το θέμα. Ως εισηγήτρια, χαίρομαι για την ανακοίνωση που είχαμε από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ζητάει μια πιο σταδιακή προσέγγιση από τη αρχική πρόταση, με την ενίσχυση της αιρεσιμότητας όσο προχωράμε από το ένα στάδιο στο άλλο. Και εκτιμώ ότι αν πρέπει να βρεθεί ένας συμβιβασμός, αυτός θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στο τρίγωνο του πότε, του ποιο θα είναι το περιεχόμενο της πρότασης, δηλαδή πόσο φιλόδοξοι θέλουμε να είμαστε μόνο ρευστότητα ή πιο πέρα, και το τρίτο, κάτω από ποιους όρους. Χρόνος, περιεχόμενο και αιρεσιμότητα. Οπότε, αν θέλετε τώρα να είσαστε πολύ φιλόδοξοι όσον αφορά το περιεχόμενο με ένα σύστημα αμοιβαιοποίησης, οι συμμετέχοντες στη συζήτηση θα πούνε ότι τότε πρέπει να αυξηθεί η μείωση του κινδύνου, που αυτό θα πάρει περισσότερο χρόνο. Αν θέλετε να ξεκινήσετε πολύ γρήγορα, πρέπει να ξεκινήσετε με την ε, ρευστοποίηση και να περιμένετε περισσότερο για την ερεσιμότητα. Οπότε μέσα σε αυτό το τρίγωνο βρίσκεται η λύση και η απάντηση. Βέβαια προς το παρόν, εδώ συγκρίνουμε μήλα μαχλάδια. Γιατί υπάρχουν εκατοντάδες διαφορετικές επιλογές στις χώρες μέλη. Υπάρχουν τόσα συστήματα διαφορετικά από χώρα σε χώρα. Και αυτή η απόκληση είναι που μας δυσκολεύει περισσότερο. Και άκουσα τον Γάλλο εκπρόσωπο που μίλησε για το γαλλικό σύστημα ότι θα στοιχήσει 7 δισεκατομμύρια παραπάνω. Ναι, αλλά τότε θα έχετε την εθνική ε, εξαίρεση και θα έχετε 0,5 αντί για 0,8. Είναι ξεκάθαρο ότι το σημείο κίνησης είναι εντελώς διαφορετικό από χώρα σε χώρα. Πάντως χαίρομαι που όλοι αναφερθήκανε στον κίνδυνο έκθεσης και στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Πάνω σε αυτά πρέπει να δουλέψουμε, εάν και εφόσον θέλουμε να προχωρέσουμε πέρα από τη ρευστοποίηση. Και κάτι άλλο, μια επιπλέον περιπλοκή είναι ότι μόνο μέρος των τραπεζών μας βρίσκεται υπό την ευρωπαϊκή εποπτεία, ενώ άλλες βρίσκονται στην εθνική εποπτεία. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Δεν θέλω να σας αποθαρρύνω, απλώς λέω πόσο περίπλοκο είναι. Και πιστεύω ότι μέσα σε αυτό το τρίγωνο κάπου θα βρούμε ένα συμβιβασμό. Ευχαριστούμε. Έστερ. Μόνο ένας μίλησε είπε ότι πρέπει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να αποτελέσουν προϋπόθεση. Αν ένας λέει κάτι που άλλοι δεν λένε, τέλο πάντων. Θα επανέλθω σε αυτό όταν πάρω το λόγο. Χρήστος Ακούρας τώρα, ΕΛΚ. Το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα έχει περάσει από διάφορα στάδια και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις. Οι τράπεζες, χώρες μέλη, υψηλά επίπεδα χρέους ιδιωτικού δημοσίου, υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι τα βασικά προβλήματα. Η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης με δύο πρώτους πυλώνες που το 2014 οι πολιτικοί προεδρία ολοκληρώθηκαν είναι ένα βασικό στοιχείο με στόχο παράλληλα να προχωρήσει και ο επιμερισμός κινδύνου και η μείωση του κινδύνου με συγκεκριμένες πολιτικές. Την ενίσχυση του εποπτικού κανονισμού και την εποπτεία ρεαλιστικά όμως με ελάχιστες κεφαλαϊκές απαιτήσει, με επίπεδα ευθύνης και με βελτίωση, όπως είπατε και εσείς, των τεχνικών διαχείρισης κινδύνου από πλευρά των τραπεζών. Χρειάζεται λοιπόν μια συνεπής αντιμετώπιση και για μείωση του κινδύνου αλλά και για την αποφυγή ε, αύξηση των ε, μη εξυπηρετούμενων δανείων και να δημιουργηθεί ένας κατάλληλος μηχανισμός και λειτουργικός ε, δικτύου προστασίας με το Ταμείο Εξυγίανσης με κατάλληλη χρηματοδότηση πρώτα και στη συνέχεια στο IMF e Και συγχρόνως να υπάρχει ένα πρόγραμμα εγγύησης ε, καταθέσεων βάσει χαρτιπορίας. Στο πρώτο στάδιο συμπληρωματικά από τα εθνικά συστήματα και στη συνέχεια με έναν μηχανισμό αμοιβαιότητας. Πιστεύουμε ότι έτσι θα μπορέσουμε να περάσουμε από την επανασφάλιση στην αποκοινού ασφάλιση. Ευχαριστώ. Βασίλεια Ηλέα, Ρουμανία. precum înființarea Fondului Monetar European. În acest sens... Ευχαριστώ. Η Ρουμανία πρέπει να σας πω ότι υιοθέτησε διάφορους νόμους και συγκεκριμένες προτάσεις Θέλουμε να συγκεντρωθούμε περισσότερο σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ των χωρών μελών δηλαδή, λαμβάνοντας όμως υπόψη τα οικονομικά συμφέροντα για την οικονομική σταθερότητα και για τη σταθερότητα των ε, δημοσιονομικών ε, της χώρας υποδοχής κάθε φορά. Το τραπεζικό σύστημα πρέπει να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να συμμετέχει στη σταθερότητα του οικονομικού συστήματος και όχι μόνο για τις χώρες της Ευρωζώνης, αλλά ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ρουμανία εκτιμά ότι είναι αναγκαίο στα πλαίσια του σχεδίου αυτού να διασφαλίσουμε ισότιμες συνθήκες για όλους και ισότιμη μεταχείριση για όλους όσοι συμμετέχουν στην ενιαία αγορά οικονομικών υπηρεσιών χωρίς διακρίσεις και χωρίς να πλήττονται τα θεμετά οικονομικά του συμφέροντα. Για τη Ρουμανία είναι πολύ σημαντική η μεταρρύθμιση του μηχανισμού ελέγχου, η εναρμόνιση των εθνικών συστημάτων εγγύησης καταθέσεων, γρήγορη αντίδραση και μηχανισμοί άπαξ και μια τράπεζα βρίσκεται σε ιδιαίτερα μεγάλη δυσκολία, μειωμένη χρήση των δημοσίων κονδυλίων για την αντιμετώπιση μιας τέτοιας κατάστασης, και επίσης σταθεροποίηση όσον αφορά την ιεράρχηση των πιστωτών. Εμείς λοιπόν συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιτευχθεί αυτό. Όσον αφορά τώρα τις αρμοδιότητες της εποπτικές και αυτό είναι κάτι το οποίο μας βρίσκει σύμφωνος. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπέρτ Λούκε από το ECR, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Μπρέκμαν δικαίως είπε ότι δεν μπορεί κανείς να χτίζει Στέγη αν δεν έχει καλά θεμέλια. Και φοβούμε ότι τα θεμέλια δεν είναι καλά όταν ε, επικεντρωνόμαστε μόνο στο AIDS και λέμε ότι το μόνο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι η μείωση και ο επιμερισμός του κινδύνου. Διότι αυτό που αγνοείται είναι ότι το έντις μπορεί να δημιουργήσει νέους κινδύνους. Ακριβώς διότι ε, μέσα ε, από ε, το σύστημα ε, ε, ε, εγγύηση των καταθέσεων θα πρέπει να κατευθύνονται σε άλλες χώρες κάτι που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο να δημιουργηθεί νέα κρίση ακριβώς επειδή θα υπάρχουν οι μηχανισμοί προστασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε δει στο παρελθόν τέτοια φαινόμενα να υπάρχει μια, μια μεταφορά του κινδύνου στις χώρες που παρέχουν τη βοήθεια και αυτό δεν αναφέρεται πουθενά στη συζήτηση, δεν αναφέρεται ούτε καν στη μελέτη επιπτώσεων της Επιτροπής, όπου δημιουργείται η εντύπωση, η εσφαλμένη, ότι το όλο ζήτημα αφορά μόνο του υπάρχοντες κινδύνους και δεν εξετάζεται καθόλου το, ο κίνδυνος να δημιουργηθούν νέοι κίνδυνοι ακριβώς μέσω αυτού του νέου συστήματος προστασίας εντό εισαγωγικών. Γνωρίζουμε ότι οι κίνδυνοι ε, που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες δεν είναι μόνο δομικοί που αφορούν τη ρευστοποίηση ή την κεφαλαιοποίηση. Πολλές φορές τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες οφείλονται στην απώλεια εμπιστοσύνης, bank run ως γνωστόν υπάρχει και αυτός ο όρος. Αυτά είναι που αποδυναμώνονται δυστυχώς ως ε, χαρακτηριστικά των τραπεζών και μέσω του ίντις και νομίζω ότι επιτέλους πρέπει να αποτελέσει θέμα συζήτηση. Ο κ. Μπαλαγούρος από την Ελλάδα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Τραπεζική Ένωση, όπως είναι γνωστό, αποτελεί ένα από τα, ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει τρεις πυλώνες. Ο πρώτος είναι η κοινή τραπεζική εποπτεία. Ο δεύτερος είναι η κοινή διαχείριση της εξυγίανσης του τραπεζών. Και ο τρίτος, ένα, δημιουργία ενός κοινού ταμείου εγγύης καταθέσεων. Στα δύο πρώτα έχουν γίνει κάποια βήματα, αλλού περισσότερο σημαντικά, αλλού λιγότερο σημαντικά και έχουν δημιουργηθεί και κάποιοι θεσμοί που υπηρετούν αυτά τα βήματα. Όμως για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα πρέπει να, να προχωρήσει το σκέλος της εγγύησης των καταθέσεων. Δεν μπορεί τα δύο μόνο να μείνουν. Χρειάζεται, ας πούμε, και το τρίτος πυλώνας. Α, υπάρχει όμως ένας πόλος μια σειρά κρατών, Γερμανίας, Ολλανδίας και άλλων, που δηλώνουν ότι πρέπει να καθυστερήσει. Η Επιτροπή μάλιστα, η Επιτροπή μάλιστα αντί να ενισχύσει τον αρχικό σχεδιασμό της, ζητά τώρα να, να εξοδετερώσουμε τους κινδύνους και μετά να ασχοληθούμε με την εγγύηση. Η ελληνική θέση μαζί με άλλα κράτη είναι υπέρ της πραγματικής τραπεζικής ένωσης που δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν διαμορφωθεί ένα αίσθημα ασφάλειας με, άμεσα, και αναγκαίο, με άμεσα και αναγκαία βήματα για την εγγύηση των καταθέσεων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you. Ευχαριστώ. Γιάννης Πούκανς από τη Λετωνία. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία αυτή που μου δίνετε να αφιερώσω δύο λεπτά να εκφράσω την άποψη της Λετωνίας για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω την υποστήριξή μου ε, για την ιδέα της ολοκλήρωσης Τραπεζικής Ένωσης. Ταυτόχρονα θα πρέπει να εισαχθούν και μέτρα για τη μείωση των κινδύνων. Πιο συγκεκριμένα, θα θέλαμε να υπάρχει υψηλότερο επίπεδο εναρμόνισης με στόχο να αυξηθεί και αποτελεσματικότητα του ενιαίου μηχανισμού. Δεύτερον, υποστηρίζουμε τη μείωση του κινδύνου ακόμα και αν χρειαστούν μεγάλες αλλαγές ε, στις νομικές ε, πράξεις που αφορούν τον τραπεζικό τομέα. Θα θέλαμε να εγκριθούν αυτές οι πράξεις ε, το συντομότερο δυνατόν και βεβαίως ε, πρέπει να βρούμε και την κατάλληλη ισορροπία στις ρυθμίσεις των τραπεζών ε, που συμμετέχουν σε διεθνείς ομίλους. Τρίτον, υποστηρίζουμε αυτό το οποίο αναφέρθηκε ήδη, το Ευρωπαϊκό ε, Μηχανισμό ε, Εγγύησης Καταθέσεων, ο οποίος θα πρέπει να συσταθεί βαθμιδών και να γίνονται πληρωμές στο σύστημα που στόχο έχουν να βελτιώσουν τη σταθερότητα του ε, τομέα. Κάτι το οποίο θα επιτρέψει να υπάρχει δημοσιονομική σταθερό, χρηματοπιστωτική συγγνώμη, σταθερότητα και να σταματήσει αυτός ο άρρηκτος δεσμός μεταξύ τραπεζών και δημοσίου χρέου. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν ωφέλη αν μπορούμε να έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα προάγει τα κρατικά ομόλογα ως ένα μέτρο σταθεροποίησης του συστήματος. Αναφέρθηκε ήδη εδώ Και εμείς βεβαίως χρειαζόμαστε μια λεπτομερή ανάλυση. Διακόπτει ο πρόεδρος, κύριε Φέλτεν, Σουηδία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η κατάσταση της χώρας της Ευρωζώνης ε, για τις τράπεζες ε, είναι πολύ διαφορετική. Έχουμε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που είναι το βασικό πρόβλημα και είναι και πολύ σημαντικός παράγον κινδύνου και νέων κινδύνων στο μέλλον. Υπάρχουν ε, πάρα πολλά προβλήματα στο τραπεζικό σύστημα και πολλές καθυστερήσεις. Ξέρω ότι χρειάζεται πολύς χρόνος για να διορθωθούν όλα τα σφάλματα τα οποία οδήγησαν στην παρούσα κατάσταση και η απάντηση του επιμερισμού κινδύνου δεν μπορεί να είναι μια ρεαλιστική λύση αν δεν επιλύσουμε ε, τα προβλήματα του παρελθόντος. Ε, η μείωση κινδύνου και ο επιμερισμό κινδύνου προφανώ και αποτελούν ικανή και αναγκαία συνθήκη. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με άλλο τρόπο. Καλό θα ήταν να ακούσουμε κάτι για τον επιμερισμό κινδύνου, για τα κόκκινα δάνεια και πώ μπορεί να γίνει αυτό ε, πριν ε, μπορέσουμε να έχουμε άρση των υπολείπων κινδύνων. Πώ μπορούμε να εμπιστευτούμε τι αγορέ για του πολίτε μα. Ο Πρόεδρο, θα πω και εγώ δύο λόγια. Καταρχάς πιστεύω ότι θα πρέπει να θυμούμαστε όλοι ότι ε, εμείς καθορίσαμε τον ενιαίο μηχανισμό εποπτείας και τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίασης. Επομένως, τώρα υπάρχει ένας επόπτης ο οποίος ε, μπορεί να δώσει επιπλέον κεφαλαϊκές απαιτήσει στις τράπεζες, να παρέμβει στη διακυβέρνηση ακόμα ε, και για τράπεζες οι οποίες είναι καθοδόν προς τη χρεοκοπία ή που κινδυνεύουν να χρεοκοπήσουν. Και φυσικά θα ήθελα να ζητήσω από όλους να λάβουν υπόψη Ποια ε, θα είναι οι χώρες οι οποίες θα μπορούν να υποφοληθούν από το ΕΝΤΙΣ ε, αν είχαν συμπεριληφθεί στη χρηματοπιστωτική κρίση. Για να συνοψίσω τώρα για τις κρατικές ενισχύσει που δόθηκαν αναχώρα. Και γνωρίζουμε επίση ότι υπάρχει το πρόβλημα του MPL, αλλά υπάρχουν και προβλήματα με άλλα στοιχεία ενεργητικού, τα οποία επίση είναι πολύ σημαντικά και ό,τι και να κάνουμε και παρεπιπτόντω υποστηρίζω το πακέτο τη Επιτροπής, το βασικό στοιχείο είναι να υπάρχει ένα επόπτη ο οποίο να είναι αποστασιοποιημένος από τα κράτη-μέλη και να μπορεί να παρέμβει εν μέρη σε, στην κατάσταση μια τράπεζα. Εκ παραλλήλου τώρα αυτό που έχουμε στα μέτρα επιμερισμού κινδύνου είναι μηδέν προ το παρόν. Και αυτό αποτελεί πρόβλημα, διότι κατά την άποψή μου το έντις δεν είναι απλώς ένα μέτρο επιμερισμού κινδύνου, αλλά είναι και ένα μέτρο μείωσης του κινδύνου. Ακριβώς ε, γιατί παρέχει κίνητρα και ε, προλαμβάνει συμπεριφορές αγοράς και καταναλωτών και προσδίδει εμπιστοσύνη στο σύστημα. Πιστεύω λοιπόν ότι αν θέλουμε να περάσουμε ε, στην ολοκλήρωση, θα πρέπει να σταματήσουμε να λέμε αμοιβαία τις διάφορες ε, ε, τυποποιημένες ιδεολογικές θέσεις και να προσπαθήσουμε να βρούμε έναν τρόπο να προσεγγίσουμε ένα τον άλλον. Οι δέσμοι μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το MPL είναι κάτι σημαντικό που μπορούμε να έχουμε και νομίζω ότι αυτό το κάναμε ως προς το, από πλευρά Κοινοβουλίου ως προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Να μην επιταχύνουμε τις διαδικασίες, να γίνουν αυτά σωστά, να δούμε ποιο είναι ο πυλώρας 2 που είναι συγκεκριμένο για την τράπεζα και την οπηλώνα σε ένα που είναι η νομοθεσία, γιατί η νομοθεσία γίνεται από τα κοινοβούλια και όχι από τον επόπτη. Χαιρετίζω λοιπόν την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί η νομοθετική πρόταση μπορεί να τελειοποιηθεί και να γίνει με έναν τρόπο που θα παρέχει τα κατάλληλα κίνητρα. Και τέλος όσον αφορά ε, ε, το δημόσιο χρέος. Ε, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η τροποποίηση, αφού η Βασιλεία αποφάσισε ότι ο κόσμος δεν θα βάλει τις τραπεζές μας σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα και δεν θα υπάρχει πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειάστηκε να αποφασίσουμε λοιπόν και αν θέλουμε να επικεντρωθούμε ακολουθώντας και τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να καθορίσουμε τα χαρακτηριστικά και, τη διαδικασία του έντις για να δούμε τι γίνεται για τη μείωση του κινδύνου και τον επιμερισμό του κινδύνου και να ξεκινήσουν κόκκινες γραμμές και φιλόδοξα σχέδια και απλώ δεν θα επιτρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ολοκληρώσει ένα σημαντικό στοιχείο του πλαισίου της Τραπεζικής Ένωσης. Πλέον επαφείται στον Ευρωπαίο νομοθέτη, αλλά νομίζω ότι και τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο και να δώσουν κατάλληλη συνεισφορά στις κυβερνήσει, διότι έχουμε ένα παράθυρο ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει χαμένο. Ο Λιβιέ, δεν ξέρω αν θέλει να πει κάτι. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να απαντήσω. Θέλουμε να ολοκληρώσουμε την Τραπεζική Ένωση, αλλά ποια Τραπεζική Ένωση. Δεν μιλάμε για την ίδια όλη, ούτε για τον ίδιο ρυθμό. Εγώ συμφωνώ με την Υπουργό πέρκε και ευχαριστώ για τη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια στο ΕΚΟΦΗΝ που εγώ ήμουν διευθυντής του Μπερνιέ. Έτσι λοιπόν πρέπει να ξέρετε ότι ναι φυσικά και πρέπει να μειωθεί ο τραπεζικός κίνδυνος και πρέπει να το κάνουμε αυτό γρήγορα για τον επιμερισμό κινδύνων επίσης. Συμφωνώ μαζί σας Πρόεδρε ότι ο επιμερισμός κινδύνου πρέπει να γίνει σε γης βάσης. Μόνο τότε θα μειωθεί ο κίνδυνος. Και όπως είπα ήδη, με το έντις δεν υπάρχει επιμερισμός κινδύνου. Πρέπει να περιμένουμε το δεύτερο στάδιο του έντις. Και λυπούμε που έφυγε η κυρία Ντελάγκη, η συγγήτρια, γιατί για την έκθεση στον κίνδυνο. Το ερώτημα είναι, θέλουμε να είμαστε ο μόνος χώρος στον κόσμο που δεν έχει μια πλήρη τραπεζική ένωση. Έτσι όπως έχει σήμερα η Ευρωζώνη δεν αποτελεί αρκετά θεμέλια. Νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε δύο φορές πριν υπονομεύσουμε τα τωρινά θεμέλια και πάμε κατευθείαν να φτιάξουμε την ε, σκεπή. πρέπει να έχουμε μια καλά λειτουργούσα τραπεζική ένωση και μετά να μπούμε στη συζήτηση για το κατά πόσο θέλουμε Λυπούμε, αλλά αν πιστεύετε ότι πρέπει να προχωρήσουμε με μηδενικό κίνδυνο, θα είμαστε μόνοι μας. Ούτε η Αμερική, ούτε η Κίνα το έχει αυτό. 27 χρόνια συζητιέται αυτό το θέμα και κανένας μεγάλος οικονομικός χώρος δεν είναι έτοιμος γι' αυτό. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι απλό Κατά τα άλλα συμφωνώ μαζί σας, Πρόεδρε. Όλα τα θέματα αυτά για την μείωση του κινδύνου είναι πράγματα που πρέπει να πάρουμε πάρα πολύ στα σοβαρά. Έχουμε μειώσει το MPL στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη κατά το 1 τρίτο τα τελευταία τρία χρόνια. Και γιατί είναι καλύτερες οι μακροοικονομικές συνθήκες. Οπότε δεν έχει να κάνει τόσο με το τι κάναμε. Το θέμα της ποσοτικής έκφρασης είναι πολύ λεπτό. Τώρα είμαστε κάτω από το 5% MPL στην Ευρωζώνη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το ζήτημα της ποσοτικής έκφρασης της μείωσης του κινδύνου δεν νομίζω ότι είναι ο σωστός τρόπος για να συζητήσουμε. Ο σωστός τρόπος είναι έχουμε ένα σύστημα για να διαχειριζόμαστε ικανοποιητικά τον κίνδυνο. Ο χάρτης πορείας του Συμβουλίου πρέπει να συμπληρωθεί με διάφορα τμήματα που να αναφέρονται στα MPLs. Πάντως η συζήτηση αυτή είναι μια σημαντική συζήτηση και μια συζήτηση που δεν μπορεί να γίνει έτσι διμερός. Συμφωνώ. Το θέμα του τι έχουμε κληρονομήσει είναι ένα ζήτημα προς συζήτηση. Τι σημαίνει και τι σημαίνει ακριβώς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 Λοιπόν,